Good afternoon, dear colleagues. Αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε παρακαλώ για να μπορέσουμε να αρχίσουμε. Η σημερινή μας συνεδρίαση θα πάει μέχρι τις 6.30 και μετά αύριο θα συνεχίσουμε από τις 9 μέχρι τις 12.30. Εφόσον δεν έχετε αντιρρήσεις σχετικά με την ημερήσια διάταξη, θεωρείται εγκεκριμένη. Ερχόμαστε τώρα στις ανακοινώσεις της Πρόεδρου. Είναι σημαντικό να ξέρετε ότι αύριο θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά 12 με 12 και 30 επί τριών θεμάτων στην ημερήσια διάταξη. Και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω λοιπόν να φέρετε τις ε, κάρτες σας για την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Και έτσι έρχομαι στο πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη που είναι εμπορική συμφωνία για την καταπολέμηση της παραποίησης απομίμησης μεταξύ αφενός Ευρωπαϊκής Ένωσης και κρατών μελών της και αφετέρου Αυστραλίας, Καναδά, Ιαπωνίας, Δημοκρατίας, Κορέας, Μεξικού και Μαρόκου, Γενέας Ιλανδίας και Σιγκαπούρης και Ελβετίας και Ηνωμένων Πολιτειών. Θα έχουμε λοιπόν μια ανταλλαγή απόψεων για το θέμα αυτό. Αλλά ίσως να θυμόσαστε κιόλα ότι ζητήθηκε από την Επιτροπή μας να γνωμοδοτήσει όσον αφορά την άκτα και τι γίνεται με τα θεμελιώδη δικαιώματα. Τώρα, ήδη από τον Φεβρουάριο η Επιτροπή είπε ότι ζήτησε την άποψη του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου όσον ε, αφορά το θέμα αυτό βάσει της συνθήκης λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τον κύριο Ντεγκούχτ είχαμε συζήτηση για αυτό το θέμα στην αρμόδια επί της ουσίας ε, Επιτροπή 29 Φεβρουαρίου στην Επιτροπή Εμπορίου και στη συνέχεια σε κάποιο εργαστήριο το Μάρτιο. Τώρα θα ανταλλάξουμε απόψεις μεταξύ μας, αφού προηγουμένως ο κ. Δρούτσας, που είναι και ο εισηγητής της Επιτροπής μας, ο συντάκτης νομοδότηση δηλαδή, για να μας ενημερώσει για την κατάσταση. Στη συνέχεια θα στραφώ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στη συνέχεια οι ευρωβουλευτές θα έχουν το λόγο. Παρακαλώ κύριε Δρούτσα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα είμαι πράγματι σύντομο, διότι πρέπει να περιμένουμε φοβάμαι έτσι και αλλιώς την απόφαση της Επιτροπής ΙΝΤΑ, της αρμόδιας επί της ουσίας Επιτροπής, για αυτό το βασικό θέμα, το κατά πόσο δηλαδή όλο, όλη αυτή η υπόθεση θα πάει τελικά για γνωμοδότηση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ή όχι. Όπως θα γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να απευθυνθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για γνωμοδότηση αλλά τώρα η Επιτροπή Ίντα, τι αυτή σκέφτεται σοβαρά την ιδέα να αποφευθεί και εκείνη εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Από ό,τι έχω καταλάβει εγώ, αύριο θα υπάρξει συζήτηση στην Επιτροπή Ίντα, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα αποφασίσουν και όλα αύριο ή όχι. Τώρα γιατί σας τα λέω όλα αυτά. Επειδή είναι ένα θέμα που πρέπει να λυθεί για να δούμε τελικά τι θα κάνει και η δικιά μας Επιτροπή ΛΥΜΠΕ με την γνωμοδότηση. Η Ολομέλεια ε, ζήτησε την άποψή μας όσον αφορά την άκτα και κατά πόσο είναι συμβατή με τις συνθήκε και κυρίως με την Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ξέρω τι τελικά θα γίνει όσον αφορά την ε, απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το κατά πόσο δηλαδή θα αποτανθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ή όχι. Εμείς μπορούμε να συνεχίσουμε τον προβληματισμό μας, αλλά να το ξεκαθαρίσω. Κατά τη γνώμη μου υπάρχουν δύο εναλλακτικές λύσεις. Από τη μια μεριά, από ό,τι φαίνεται, έχουμε την τελική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αποτανθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για γνωμοδότηση δεν ξέρουμε κατά πόσο θα κάνει το ίδιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφασίσει να αποτανθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και αυτό, τότε, σύμφωνα με τον κανονισμό μας, αλλά εδώ θέλω και η Γραμματεία να με βοηθήσει και να μας πει τι ακριβώς ισχύει, τότε λοιπόν οι διαδικασίες όσον αφορά τις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές σταματούν, μπλοκάρονται. Τώρα, πολιτικά μιλώντα, εφόσον και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτοθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για το ίδιο θέμα, τότε αναρωτιέμαι πώ εμεί ω Επιτροπή ΛΥΜΠΕ μπορούμε νομικά να ασχοληθούμε με το θέμα τη άκτα. Γιατί δεν νομίζω ότι θα ήταν σόφρον να μπούμε σε ανταγωνισμό κατά κάποιο τρόπο με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σε νομικού όρους. Αυτά λοιπόν είχα να καταθέσω εδώ και θα ήθελα να ακούσω και τους συναδέρφους ποια είναι η γνώμη τους, πώς νομίζουν ότι πρέπει να προχωρήσουμε, τι διαδικασία να ακολουθήσουμε. Περιμένοντας βέβαια έτσι καλώς να δούμε τι θα κάνει και η Επιτροπή ΙΝΤΑ εσωτερικού εμπορίου. Αυτές είναι οι πρώτες μου σκέψεις εισαγωγικά όσον αφορά τη διαδικασία. Αν δεν λυθεί το διαδικαστικό ζήτημα, φοβάμαι ότι δεν θα είμαστε σε θέση να μπούμε και στην ουσία του ζητήματος. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κύριε Δρούτσα. Να ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρώτα. Κύριος Αντρεσγέσεν, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ μπορώ πολύ σύντομα να σας ενημερώσω πώς έχει η κατάσταση από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όσον αφορά τη γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, όντω, οι Νομικέ υπηρεσίε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχουν ξεκινήσει διαβούλευση μεταξύ των υπηρεσιών μα ε, προκειμένου στι 20 Μαρτίου, στην προθεσμία δηλαδή των 10 ημερών, μάλλον μετά από τις 20 10 μέρες, ε, έχουμε εργάσιμες που πάμε δηλαδή 10 Απριλίου προκειμένου να ε, πάρουμε την απόφαση, που σημαίνει ότι έτσι θα φτάσουμε στα τέλη Απριλίου. Εφόσον βέβαια χρησιμοποιήσουμε τον ε, αναγκαίο μόνο χρόνο, τον ελάχιστο αναγκαίο χρόνο. Αυτά για την γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Τώρα όσον αφορά τα κράτη-μέλη. Και σε σχέση με αυτά που είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο εργαστήριο της ΙΝΤΑ. Ε, Μια μικρή αλλαγή υπάρχει από την Κύπρο, γιατί η Κύπρος σκοπεύει να υπογράψει και εκείνη. Πότε ακριβώς δεν ξέρουμε. Όσον αφορά πάντως στις άλλες χώρες μέλη, δεν υπάρχουν αλλαγές. Η κατάσταση παραμένει όσοι είχε και σε εκείνη τη συνάντηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Γένσεν, λέει πρόεδρος. Συζήτηση τώρα. Οι συνάδελφοι. Η Ρενάτα Βέμπερ έχει ζητήσει πρώτα το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Αναμφισβήτητα η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για να ε, ε, αποδεχθεί ή να απορρίψει τη συμφωνία θα είναι μια πολιτική απόφαση. Γι' αυτό και τώρα είμαστε σε κάποια στιγμή όπου έχουμε τα κράτη-μέλη τα οποία αρχικώς είχαν ε, υπογράψει τη συμφωνία τώρα θέλουν να αποσύρουν την υπογραφή ή άλλαξαν γνώμη διότι ε, δυστυχώς ε, υπέγραψαν κάτι χωρίς να ξέρουν καν τι υπέγραψαν. Και όταν κοιτάζει κανείς ε, τις σχέσεις ε, μεταξύ κυβερνήσεως και πολιτών βλέπουμε ότι υπάρχουν προβλήματα. Επίσης ε, ε, όταν έχουμε μόνο μία γνωμοδότηση σαν ε, ανηλυμένη ευθύνη της Επιτροπής Ελευθεριών είναι ατυχές διότι τα θέματα δεν είναι μόνο για την Επιτροπή Ίντα αλλά και η οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελευθεριών. Το ερώτημα λοιπόν είναι τι ρόλο θέλει να παίξει, πόσο ο δραστήριος σκοπεύει να είναι ε, όσον αφορά την παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο διότι θα είναι πολιτική ψηφοφορία και το ε, τονίζω. Πρέπει λοιπόν να θέσουμε προς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο τις ερωτήσεις. Ε, εδώ δεν μιλάμε για την άποψή του την οποία ζητούμε και είναι σημαντικό να μπορέσουμε να λάβουμε τη σωστή απάντηση και από πλευράς νομικής. Όσον αφορά την παραπομπή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αντιλαμβάνομαι ότι θα είναι σε πολύ γενικές γραμμές. Δηλαδή, ε, στην πολιτική μας ομάδα συζητήσαμε το θέμα με την Επιτροπή Ίντα και λέχθη ότι θα έπρεπε να τεθούν περισσότερα ερωτήματα ε, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Οπότε εγώ επιμένω ε, ότι η Επιτροπή Ελευθεριών πρέπει να παίξει ένα πιο ουσιαστικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία και χωρίς ε, να, ε, να κάνω έκκληση τουλάχιστον ενθαρρύνω τον εισηγητή μας να παραπέμψει ε, τα θέματα αυτά ή στην ΙΝΤΑ διότι ε, θα πρέπει ε, να μπορούμε να εκφραστούμε και είναι βασικό να μπορέσουμε κατ' εμέ που είμαι υπέρ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να παραπέμψει το θέμα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και όχι σε γενικές γραμμές αλλά με πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα και αυτό να περιλαμβάνει και όλες τις ε, νομικές πτυχές που απασχολούν τα κράτη-μέλη που πρόκειται να εφαρμόσουν αυτή την εφαρμογή. Ευχαριστώ κύριο Σλάιτερ. Και εγώ ήμουν προηγουμένως στην Επιτροπή ΙΝΤΑ και παρακολουθώ αυτή τη συμφωνία εδώ και χρόνια. Στην αρχή έπρεπε να είχαμε δυσκολία να έχουμε πρόσβαση και στην πληροφόρηση, αλλά τώρα την παρακολουθούμε εδώ και χρόνια. Από την αρχή Είχαμε ανησυχήσει για τον περιορισμό των δικαιωμάτων μας και τώρα που άλλαξα επιτροπή θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει ενισχυμένη συνεργασία διότι η συμφωνία ΑΚΤΑ δεν αναφέρεται μόνο στα ανθρώπινα δικαιώματα αλλά σε διάφορα θέματα και συμφωνώ απολύτως με αυτά τα οποία μόλις ελέγχθησαν. Θα ήθελα όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην διότι ε, αντιλαμβάνομαι ότι αρχές Απριλίου θα έχει ολοκληρωθεί η συζήτηση μεταξύ των υπηρεσιών. Ε, είσαστε όμως βέβαιοι ότι από εκεί και πέρα θα υπάρξει ε, μία δέσμευση από την Επιτροπή Πολιτική η οποία θα εξασφαλίσει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προχωρήσει και θα προχωρήσουν στην παραπομπή δεν ξέρουν πώς θα διαμορφώσει ερωτήσεις θα μπορούσε το Κοινοβούλιο να διατυπώσει μόνο του ερωτήσεις και παραδείγματο χάρη διαφορά τιμών. Θα ήθελα λοιπόν να έχουμε ε, απαντήσεις στις ερωτήσεις μας βάσει των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μην είμαστε εκ των υστέρων δυσαρεστημένοι με τις ερωτήσεις που θα θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θεωρούμε όμως ότι το να παραπέμψει το θέμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η λογική συνέχεια και αυτό όμως ε, ε, δεν είναι προφανές ότι ε, το δικαστήριο θα αποφασίσει υπέρ ημών διότι μπορεί πολιτικά να μην είναι σωστό και το δικαστήριο να λάβει άλλη νομική απόφαση οπότε εμείς θα πρέπει να διατυπώσουμε δικές μας ερωτήσεις και να δούμε ποια είναι η αξία των συμφωνιών αυτών από πλευράς ανθρωπίνων δικαιωμάτων διότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να προχωρήσει μπορεί να έχουμε απλώς ακροάσεις ή ε, ε, βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλές ενδιαφέρουσες απόψεις από την διακήρυξη του Ανοβέρου ε, υπάρχει επίσης μία αξιολόγηση της ΣΑΚΤΑ και από επίπεδο πολιτικής θα πρότεινα να έχουμε ένα έγγραφο σαν αυτό αλλά να αναφέρεται στην ε, Συμφωνία Άκτα. Οπότε ήδη από τώρα ανεξαρτήτως από την ε, έκβαση της ε, ερωτήσεως στο Κοινοβούλιο θα μπορούσαμε και εμείς να διατυπώσουμε την, τη δικιά μας κρίση. Ευχαριστώ, κύριος Μπουζουτήλ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πιστεύω ότι αν, για, αν και πρόκειται για μια εμπορική συμφωνία, τα ζητήματα που θίγει κινούνται πέραν της εμπορικής συμφωνίας. Μιλάμε για πολιτικές ελευθερίες. Διάβασα αυτή τη συμφωνία από, και αν έπρεπε να τη διαβάσω από εμπορική σκοπιά, δεν θα είχα να αντιτάξω κάτι, αλλά υπάρχουν πολλά ερωτηματικά σε σχέση με τις πολιτικές ελευθερίες και κατά πόσο υπάρχουν δυσανάλογοι περιορισμοί στη... ναι, στις ελευθερίες ως προς τη ε, χρήση του διαδικτύου. Και πολλοί έθεσαν παρόμοια ερωτήματα. Τώρα εμείς τι ρόλο, ποιο ρόλο μπορούμε να διαδραματίσουμε επί του θέματος. Όπως είπε η κυρία Βέμπερ, δεν θα ήθελα να γίνει προσφυγή στο ΔΕΚ. Δεν θα ήθελα να αποστείλει μια επερώτηση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αν γίνει όμως το θέμα, τότε θα πρέπει να σταματήσουμε να το συζητούμε μέχρι ότου αποφανθεί το δικαστήριο. Χρήζει όμως συζήτησης, διότι υπάρχει μεγάλη παραπληροφόρηση επί του θέματος και πολλοί προσδοκούν από μας να απαντήσουμε σε αυτά τα ερωτήματα και να συζητήσουμε την άκτα, την εμπορική συμφωνία αυτή από πλευράς πολιτικών ελευθεριών. Ακόμα και αν ε, προσφύγουμε στο ΔΕΚ, θα πρέπει ως Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών να μην σταματήσουμε τις συζητήσεις επί του θέματος. Καλωσορίζω λοιπόν το θέμα ότι σήμερα έχει ενταχθεί στην ημερήσια διάταξη το θέμα προς συζήτηση και θα ήθελα να παραμείνει έτσι ώστε να συνεχίσουμε να το συζητάμε το θέμα αναμένοντας και αποφάσεις από την Κομισιόν και απαντήσει από την Κομισιόν. Θα ήταν σκόπιμο να συμμετάσχουμε ενεργά στις συζητήσεις της ΙΝΤΑ. Το προτρέπω και τον εισηγητή για το ίδιο. Οι συζητήσεις άρχισαν κατά τα τέλη Φεβρουαρίου και γι' αυτό θα πρέπει να εισακουστεί και η άποψη της ΛΥΜΠΕ ως προς την οπτική γωνία των πολιτικών ελευθεριών. Θα πρέπει να διασαφινιστεί το ζήτημα και δεν νομίζω ότι οι διαπραγματευτές ήθελαν να περιστήλουν τις πολιτικές ελευθερίες και την ελευθερία χρήσης του διαδικτύου. Εάν όμως αυτές ήταν οι προθέσεις θα πρέπει να το γνωρίζουμε έτσι ώστε να έχουμε μια πλήρη πληροφόρηση και να συμφωνήσουμε ή όχι με την συμφωνία. Η κυρία Ιντφέλτ. Συμφωνώ ότι μιλάμε για ε, νομικές, ε, νομικές συμβουλές και πολιτικού χαρακτήρα συμβουλές. Αυτό όμως δεν σημαίνει εξωτερική ανάθεση του ζήτηματος. Εάν υπάρχουν πραγματικές αμφισημίες που δεν μπορούμε να αποσαφηνίσουμε με τη δική μας νομική υπηρεσία ή την αντίστοιχη της Επιτροπής ή τον Οργανισμό Θεμελιωδών Ελευθεριών, γιατί από εκεί αρχίζουν οι αντιρρήσεις ως προς την άκτα, τότε να προσφύγουμε στο ΔΕΚ. Αλλά αυτή είναι και η τελευταία μας επιλογή. Και ο Σάιμον Μπουζούτιλ πολύ σωστά είπε ότι ελοχεύει ένας κίνδυνος Δηλαδή θα παραλύσει η όλη συζήτηση. Τουλάχιστον ας ζητήσουμε τη νομική αρρωγή αυτών των οργανισμών και υπηρεσιών και όπως ξέρετε αύριο θα ψηφίσουμε το PNR, δηλαδή τα προσωπικά δεδομένα επιβατών, όπου δεν ζητήσαμε την γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας και θα προσφύγουμε παρόλα αυτά στο ΔΕΚ. Άρα υπάρχει μία αντίφαση εδώ. Υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο, γιατί πρόκειται για κάτι που μπορούμε να κάνουμε και εμείς οι ίδιοι. Δηλαδή να υπάρχει πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα ως προς τις διαπραγματεύσεις. Αυτό το προώθησα το 2008 όταν πρωτοσυζητήσαμε το θέμα. Ο εισηγητής φαίνεται ότι είναι κάπως αφηρημένος ή απασχολημένος. Εν πάση περιπτώσει, προέβαλα ένα αίτημα και ζήτησα την σχετική τεκμηρίωση. Προσέφυγα στο ΔΕΚ που συζητά το θέμα το έθιξα και πριν από 1,5 μήνα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε ότι τα πρακτικά που αφορούν τους προηγούμενους γύρους διαπραγματεύσεων θα μπορούσαν να διαβιβαστούν. Αλλά πολλά πρακτικά δεν είναι ευανάγνωστα. Και ο ε, υπάλληλος που μου απέστειλε το κείμενο, αντί να διαγράψει αυτά που έπρεπε να διαγράψει, τα τόνισε, τα υπογράμισε. άρα μάθαμε αυτά που δεν θα έπρεπε να γνωρίσουμε. Εν πάση περιπτώσει, δεν το κοινοποίησα στην ιστοσελίδα μου, αλλά θα μπορούσα να σας κοινοποιήσω αυτά τα στοιχεία, αν το επιθυμείτε, αφού έγινε αυτό το λάθος. Όχι τώρα μιλώντας σοβαρά για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, ειδικά αυτά που είπε ο Σάιμον, δηλαδή να γνωρίζουμε τις προθέσεις των διαπραγματευτών, που γνωρίζουμε πολύ καλά πλέον. Βεβαίως η Επιτροπή μας είπε ότι δεν μας ενδιαφέρουν μόνο οι προθέσεις, αλλά νομίζω ότι ένα από τα στοιχεία κλειδιά είναι πώς θα ερμηνευτεί αυτή η συμφωνία έμπρακτα. Αυτή είναι μία από τις βασικές αμφισημίες, διότι η Κομισιόν μας μιλά για εφαρμογή της προϋπάρχουσας νομοθεσίας, ενώ όσοι αντιτάσσονται αναφέρουν ότι πρέπει να δημιουργηθεί νέα νομοθεσία. Αυτό είναι το θέμα καθαρά ερμηνείας και προθέσεων. Και νομίζω ότι η Επιτροπή μας και ο εισηγητής θα πρέπει να έχουμε πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με τις διαπραγματεύσεις, έτσι ώστε να έχουμε τη δική μας γνώμη σε σχέση με τις προθέσεις και πώς θα πρέπει να ερμηνευτούν όλα αυτά. Και τέλος, είδα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάπως ενοχλήθηκε γιατί προβλήθηκε μια εκστρατεία κατά της άκτα και είπε ότι ότι δεν μπορούμε να ακούμε τις φωνές που προέρχονται από τους δρόμους. Μα αυτό δεν ενθαρρύνουμε ακριβώς στις ε, χώρες του αραβικού κόσμου. Και οι νέοι και στην Ευρώπη οργανώνονται και προβάλλουν εκστρατείες. Αυτό δεν θέλουμε τη συμμετοχή των ανθρώπων και δι των νέων στην πολιτική. Ο κύριος Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εντάχει, καταρχήν να ευχαριστήσω τον κύριο Δρούτσα που έχει ενώπιόν του ένα αμφίσιμο ζήτημα. Θα ήθελα να πω ότι με κάλυψε ιδιαίτερα ο κύριος Μπουζούτιλ και να προσθέσω ότι φυσικά θα πρέπει να προστατεύσουμε τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών, αλλά από το ηλεκτρονικό μου ταχυδρομείο βλέπω τη μία πλευρά του θέματος. Τι σημαίνει η άκτα. Θα πρέπει να δούμε και τις θετικές πτυχές της εμπορικής αυτής συμφωνίας κατά πολέμησης της παραποίησης. και την προστασία εκείνων που είναι δημιουργοί και που θα πρέπει ελεύθερα να διαδίδουν και να διανέμουν αυτά που δημιουργούν. Θα ήθελα να σας, ε, ε, να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία, να φτάσετε σε μία εξισορρόπηση και ελπίζω το ΔΕΚ να ρίξει κάποιο φως στο όλο ζήτημα. Σας ευχαριστώ και καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε τον κύριο Παπα-Νικολά, κυρία Φάιλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καιρός είναι που συζητάμε σήμερα την άκτα Δυστυχώς είναι κάπως άδεια η αίθουσα για μια τόσο σημαντική συζήτηση, ιδιαίτερα αν λάβουμε υπόψη μας πως οι πολίτες τις τελευταίες εβδομάδες έδειξαν ότι περιμένουν τη δικιά μας την αντίδραση. Παραμένουν πολλά ανοιχτά ερωτήματα από ό,τι φαίνεται για τη συνέχεια της διαδικασίας. Θέλω όμω να υπογραμμίσω εδώ ότι υπάρχει μια προφορική ερώτηση δικιά μου και άλλων πέντε συναδέλφων προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και μια που είναι εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ίσω ήδη να μπορεί να δώσει κάποιε απαντήσει για την επικύρωση τη άκτα. Λαμβάνοντα υπόψη ότι υπεγράφει από 22 χώρε μέλη, ότι αντιτίθεται οι πολίτες και τους στηρίζουν και διάφοροι ειδικοί της κοινωνίας των πολιτών, μη κυβερνητικών οργανώσεων κλπ. Θα ήθελα να γνωρίζω τι θα γίνει εάν ο αριθμός των χωρών μελών ε, δεν είναι πλησάν, δηλαδή δεν επικυρώσουν όλες οι χώρες. Και ποιες θα ήταν οι επιπτώσεις της μη επικύρωσης κάποιων ε, ατομικά χωρών μελών. Εδώ παραμένουν κάποιες αβεβαιότητες και καλό θα ήταν να δοθούν απαντήσεις πριν αρχίσουμε να συζητάμε στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές. Γιατί ίσως ολόκληρο το εγχείρημα, η ψηφοφορία κτλ. να μην λάβουν ποτέ χώρα. Τώρα, όσον αφορά την παραπομπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για το θέμα αυτό. Όντως θα καθυστερήσει την όλη διαδικασία και σημαίνει ότι στο μεταξύ θα σταματήσει η όλη συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γι' αυτό λοιπόν είμαι πολύ διστακτική και το είπα αυτό και στην ομάδα μου όταν το συζητήσαμε. Το ίδιο ισχύει και για την προσωρινή έκθεση που προτείνει ο εισηγητής της Επιτροπής ΙΝΤΑ. Έχω κάποιες αφιβολίες βλέπετε κατά πόσο θα βοηθήσει μια τέτοια διάμεση έκθεση, γιατί η έκθεση έχει συζητηθεί και το μόνο που μένει είναι να πούμε ναι ή όχι. Μήπως πάλι πρόκειται μόνο για καθυστέρηση της διαδικασίας. Εννοείται ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη συμφωνία. Το όλο αυτό θέμα όμως πρέπει να το δούμε και πολιτικά, όχι μόνο νομικά. Ο Σάιμον αναφέρθηκε σε πολλά σημεία. Είπε πολλά επιχειρήματα γιατί δεν πρέπει να επικυρωθεί η άκτα, γιατί πρέπει να καταψηφιστεί. Δεν θα πω εγώ τώρα στο περιεχόμενο, στην ουσία. Θα υπογραμμίσω όμως κάποια πράγματα και μερικά από τα επιχειρήματά του. Μερικές μεγάλες χώρες δεν υπογράφουν Συνεπώς, η άκτα είναι το κατάλληλο εργαλείο για να καταπολεμήσουμε την παραπίση και την απομίμηση. Δεν νομίζω. Από την άλλη άκτα δεν είναι μια διεθνής σύμβαση. Και έτσι οι διαπραγματεύσεις έγιναν με μυστικότητα. Έπειτα η συζήτηση για το copyright στο διαδίκτυο, τα βασικά δικαιώματα, οι ελευθερίες είναι πράγματα που πρέπει να συζητιώνται δημόσια, ανοιχτά, στα κοινοβούλια, κάτι το οποίο δεν έγινε. Και έχουμε και την αίσθηση ότι υπάρχει πίεση από την αμερικανική βιομηχανία, τουλάχιστον εγώ έχω αυτή την εντύπωση. Επίσης, ε, τα πράγματα πάνε γρήγορα και οι ερμηνείες που δίνονται είναι πολλές και διάφορες για την άκτα. Ακόμα κι αν δεν λέει πουθενά ότι υπάρχει λογοκρισία στο διαδίκτυο, παρόλα αυτά η άκτα έχει μια τέτοια τάση περιορισμού της ελευθερίας και μπορεί να δημιουργήσει μεγάλες αλλαγές στην προστασία των δεδομένων. Έπειτα κάτι άλλο πολύ σημαντικό είναι το θέμα της πνευματικής ιδιοκτησίας. Κατά πόσο με την άκτα ε, λύνουμε αυτό το ζήτημα δεν ξέρω. Πρέπει πιστεύω να συζητήσουμε περισσότερο για τη δημοκρατία και ίσως να έχουμε ένα νέο κανόνα για την πνευματική ιδιοκτησία και να μην καλύπτεται από την άκτα. Πιστεύω λοιπόν ότι χρειάζεται περισσότερο πολιτική συζήτηση. Οπότε από αυτή την οπτική γωνία χαίρομαι που στις 12 Απριλίου θα γίνει συζήτηση για αυτό το θέμα με εκπροσώπους όλων των μερών. Η αντίθεση των πολιτών για μένα αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία να συζητήσουμε δημόσια τη συμφωνία και μόνον αφού έχουμε συζητήσει και δούμε ότι η κοινωνία των ε, πολιτών θέλει και ότι οι εμπειρογνώμονες λένε ναι, μόνο τότε να μπορούμε και εμείς να εγκρίνουμε. Και συμφωνώ και με αυτό που είπε και η Σόφη, ότι εμείς ως Κοινοβουλευτική Επιτροπή πρέπει να ζητήσουμε ελεύθερη πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα τα οποία ήδη υπάρχουν και έχουν να κάνουν με τη Συμφωνία Άκτα. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ο κύριος Άντζο έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν έχω να προσθέσω και πολλά. Άκουσα από τους συναδέλφους όλα όσα μπορούν να λεχθούν σε σχέση με αυτό το θέμα. Θα ήθελα να προσθέσω μόνο ένα στοιχείο. Αποδεικνύεται για άλλη μία φορά ότι όσοι θεωρούν ότι μπορούν να αποφασίσουν ένα θέμα και να το θεωρήσουν θέμα απόρριτο, κάνουν ένα πολύ μεγάλο λάθος. Δεν μπορεί να αποφασιστεί με μυστικότητα. Και γι' αυτό ακριβώς είχαμε μεγάλη παραπληροφόρηση και ιδιαίτερα του κοινού. Όπως είπε πολύ σωστά και η κυρία Ιντβέλτ, καταρχήν θα πρέπει να ακούσουμε τις φωνές που προέρχονται από τους δρόμους από το κοινό, από τους νέους. Να δούμε αυτή την αρνητική πτυχή που αφορά την άκτα και τη χρήση του διαδικτύου. Θα πρέπει να προστατεύσουμε τους νέους, να προβάλλουμε την δημιουργικότητα. Νομίζω ότι ο εισηγητής μας θα πρέπει στις προσεχείς διαπραγματεύσεις να διατρανώσει τη θέση μας, γιατί όπως είπαν οι συνάδελφοι, δεν μιλάμε για εμπορική συμφωνία, δεν μιλάμε για το εμπορικό σκέλος της συμφωνίας, αλλά για το σκέλος των πολιτικών ελευθεριών, ιδιαίτερα μέσω διαδικτύου. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να δράσουμε πιο συνεκτικά και με σπουδή. γιατί δεν θα υπάρξει εύκολη συνεννόηση με τα κράτη-μέλη και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν ξέρω γιατί. δεν ξέρω, δεν νομίζω πάντως ότι θα είναι εύκολη η συνεννόηση. Πριν δώσω το λόγο στον εισηγητή, θα ήθελα να ρωτήσω την Επιτροπή κατά πόσο θέλει να απαντήσει στα ερωτήματα που υποβλήθηκαν. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, ελπίζω ότι πήρα όλες τις ερωτήσεις, έχω σημειώσει όλες τις ερωτήσεις. Καταρχήν το ο, θέμα της παραπομπής. Όπως ελέγχθη, ε, το Συμβούλιο, το Κολέγιο των Επιτρόπων αποφάσισε να γίνει αυτή η παραπομπή στο δικαστήριο και το θέμα είναι πότε ακριβώς θα υιοθετηθεί το ερωτηματολόγιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά εντός του Απριλίου φαντάζομαι ότι θα προχωρήσουμε και η νομική υπηρεσία κινείται τώρα βάσει αυτής της αποφάσεως. Δεύτερον, σχετικά με το τι συμβαίνει εάν κάποιο άλλο κράτος μέλος δεν υπογράψει, τελικά αν δεν ε, υπογράψουν αρκετά κράτη τότε δεν θα μπορέσει να υπάρξει συμφωνία και αυτό είναι σαφές. Και σε προηγούμενα θέματα, ε, δεν ξέρω σε τι θέμα αναφερόταν ε, ο κύριος Ευρωβουλευτής, αλλά γενικώ έχουμε ζητήσει, έχουμε θέσει τις ερωτήσεις αυτές και στο παρελθόν και από εκεί και πέρα άπαξ και τα κράτη-μέλη δεν υπογράψουν, τα κράτη που απεφάσισαν ε, μόνο προσφάτως ε, στο Συμβούλιο ή σαν μέλη του Συμβουλίου να ψηφίσουν ε, ενδέχεται να υπάρξουν 22 κράτη τα οποία ήδη έχουν αποφασίσει να υπογράψουν και που δεν είναι λόγο δεν εμποδίζει το γεγονός ότι κάποιος ε, δεν ε, υπογράφει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ε, διατυπώσει τις δικές του απόψεις. Δεν θα αναφερθώ τώρα εις ε, το θέμα το οποίο εκρεμεί στο δικαστήριο σχετικά με την πρόσβαση στα έγγραφα και θα επαναλάβω αυτό που έχει λεχθεί γενικώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του θέματος ότι ναι τα έγγραφα αυτά είναι σημαντικά αλλά είναι πολύ βασικό να δούμε τι λέει το τελικό κείμενο και ε, ορισμένα σχόλια αναφερόντουσαν στα έγγραφα τα οποία δεν περιλαμβανόντουσαν στη συμφωνία είτε διότι δεν συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις ή γιατί το τμήμα αυτό των διαπραγματεύσεων είχε απορριφθεί από τους άλλους συμβαλόμενους. Είναι ε, δύσκολο λοιπόν να πούμε ότι όποιο ο κείμενο δεν, ε, ε, δεν έγινε αποδεκτό, θα ε, συμπεριληφθεί στο τελικό κείμενο. Θέλω να διευκρινίσω, εγώ μιλώ για έγγραφα τα οποία δεν διέρευσαν, μου τα έστειλαν επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και απλώς το λάθος που έγινε ήταν ότι ορισμένα σημεία είχαν διαγραφεί. Δεν είχαν διαρρεύσει όμως και υποθέτω ότι μπορώ να τα δείξω σε οποιοδήποτε ε, ενδιαφέρεται, εφόσον δεν πρόκειται για διαρροή. Ο κύριος Γιάννησεν. Θέλω να διευκρινίσω και σας είπα ότι δεν θα σχολιάσω τη συγκεκριμένη περίπτωση, απλούστατα αναφέρομαι γενικώ στα έγγραφα τα οποία κυκλοφορούν στα blogs. Γι' αυτά που στάλησαν σε εσά είναι ένα θέμα που εκρεμεί αυτή τη στιγμή. Ο κύριος Δρούτσας έχει τώρα το λόγο για να κλείσει. Ευχαριστώ και ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για τα σχόλια και τις σκέψεις που εξέφρασαν όπως άλλωστε και τις ε, προτάσεις. Βεβαίως συμφωνώ ότι είναι ένα πολύ πολιτικοποιημένο θέμα το και θα πρέπει να υπάρξει μία πολιτική συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Η ε, δραστήρια συμμετοχή της Επιτροπής Ελευθεριών και μου προσωπικά ως ε, εισηγητή μου φαίνεται ε, ε, σαφής ε, και προφανής. Ε, επίσης χαίρομαι που υπάρχουν αυτά τα διάφορα σχόλια από συναδέλφους και ότι υπάρχει μία στήριξη για αυτή την ενεργή συμμετοχή. Και λυπούμε που εκφράζομαι έτσι, αλλά δεν ξέρω πώς θα το... Θα το προωθήσω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι η επίσημη επιτροπή είναι η ΙΝΤΑ. Πρέπει να δούμε λοιπόν πώς θα αντιμετωπίσουμε τις συζητήσεις και πώς θα συνεργαστούμε με την Επιτροπή ΙΝΤΑ. Επίσης, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Επιτροπή Ελευθεριών έχει αναλάβει από την ε, Ολομέλεια να εξετάσει την συμβατότητα με τα δικαιώματα τα οποία περιλαμβάνονται ε, στον ε, χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων, δηλαδή να συγκρίνει την άκτα με αυτό το χάρτη. Και θεωρώ ότι ήταν βασικό στην πρώτη μου παρέμβαση να θέσω ορισμένα διαδικαστικά ερωτήματα. Πρέπει να διευκρινίσουμε το σημείο αυτό, αλλά πρέπει να σας πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερος ακούγοντας τους συναδέλφους ότι ερμηνεύουμε ε, την ε, εντολή που έχει δοθεί στην ε, Επιτροπή Ίντα ως ευρεία και μπορώ να αποδεχθώ ευχαρίστως ε, αυτή την πρόταση και ε, θα αναλάβουμε αυτή την δέσμευση. Γι' αυτό και προτείνω διαδικαστικά να ζητήσω από τους συναδέλφους που είναι σκιώδεις να συναντηθούμε αμέσως δηλαδή στα πλαίσια αυτής της εβδομάδος στις Βρυξέλλες και να δούμε πώς θα συνεχίσουμε την εργασία μας, πώς θα οργανωθούμε μετά από αυτή την ε, ανταλλαγή απόψεων και να σας πω ότι είναι για μένα αυτονόητο όχι μόνο διότι αυτό είναι ένα θέμα και μία πτυχή της άκτα που είναι πολύ σημαντική και πολύ πολιτικοποιημένη και ε, πολύ ενδιαφέρουσα για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες και γι' αυτό σας εγγυώμαι ότι ε, θα υπάρξει πλήρη συνεργασία με όλους τους συναδέλφους από όλες τις πολιτικές ομάδες και θα ολοκληρώσω αναφερόμενος στο ε, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και τις ερωτήσεις που θέλει να απευθύνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εγώ ε, αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν ορισμένα προβλήματα στο να προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση διότι εφόσον έχουμε την Επιτροπή η οποία ούτως ή άλλως θα προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εάν το πράξει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ε, ε, δημιουργήσουμε την εντύπωση στην κοινή γνώμη ότι προσπαθεί να καθυστερήσει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με όλο το σεβασμό προς τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εάν παραπέμψουμε το θέμα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα δώσουμε πολιτική κάλυψη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στον τρόπο με τον οποίο έχει διεξάγει τις διαπραγματεύσεις επί της άκτα μέχρι ότου ολοκληρωθούν. Βέβαια πρέπει να δούμε ε, τι θα είναι οι παραπεπτικές ερωτήσεις τις οποίες θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και αυτό θα ήταν το πιο φρόνιμο εξού και δέχομαι την πρόταση της κυρίας Σίντφερτ. ε, με συγχωρείτε που σας διέκοψα αλλά θέλω να σας πω ότι συμφωνώ με την άποψή σας ότι θα πρέπει να στραφούμε προς τις υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να προσπαθήσουμε να ε, διευκρινίσουμε όλα αυτά τα θέματα και να δούμε τι ερωτήσεις πρέπει να απευθύνει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αν αποφασίσει να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση και επιπλέον να ζητήσουμε και να απαιτήσουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να, λάβει, να ε, έχει πλήρη πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα. Αν όλοι λοιπόν συμφωνήσουμε, ο καλύτερος τρόπος είναι να συναντηθούμε μέσα στις επόμενες ημέρες και αύριο αν είναι δυνατόν και αν έχουν ελεύθερο χρόνο όλοι οι σκιώδεις εισηγητές για να γίνει αυτή η πρώτη ανταλλαγή απόψεων, να δούμε πώς θα οργανωθούμε, πώς θα συνεχίσουμε, άπαξ και η Επιτροπή Ελευθεριών έχει εκφράσει την θέληση και την δέσμευση ότι ο ρόλος του Κοινοβουλίου δεν περιορίζεται εις ε, την ε, μετά δοσημιάς γνωμοδοτήσεως αλλά σε μια ευρύτερη ε, συζήτηση. Ευχαριστώ. Ε, κύριε Σλάιτερ, θέλετε να συζητήσετε μετά την κυβέρνηση, μετά τη συνεδρίαση την ερώτησή σας προς τον κύριο Δρούτσα. Ευχαριστώ. Μήπως ε, ήταν στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η παραπομπή αυτή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αλλά από τη δικιά μας την ε, πλευρά, τι θα γίνει αν η ΙΝΤΑ συνεχίζει τις δικές της διαδικασίες και η δικιά μας η αξιολόγηση βάσει του άρθρου 36 αν είναι ανεξάρτητα από την απόφαση του δικαστηρίου, γιατί εκείνες ασχολούνται με το κατά πόσο είναι συμβατό το θέμα με τις συνθήκες. Ενώ αν η δικιά μας άποψη είναι ότι πρόκειται για κάτι ασύμβατο με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τότε ποιο είναι το νομικό καθεστώς μιας τέτοιας γνωμοδότησης. Τι σημαίνει. Σημαίνει ότι εμείς θα ψηφίσουμε όχι, δεν θα δώσουμε σύμφωνη γνώμη. Δηλαδή, τι σημαίνει ακριβώς αυτή η γνωμοδότηση στην πραγματικότητα. Για να ξέρω δηλαδή όταν συναντηθούμε τι ισχύει, να το ξέρω από πριν για να δω τι θα κάνω στη συνάντηση αυτή. Να το ρωτήσετε ίσως με τους συντονιστές ή έχετε απάντηση κύριε Δρούτσα. Δυστυχώς δεν είμαι σε θέση να απαντήσω. Όντως ήταν και ένα από τα πρώτα μου ερωτήματα ακριβώς. Προτείνω λοιπόν εντελώ πρακτικά να προσκαλέσουμε και την γραμματεία να έρθει στην συνάντησή μας αυτή αύριο μεθαύριο όποτε γίνει και να δούμε μήπως ε, γίνεται να προετοιμαστεί η γραμματεία για να έχει κάποιες απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά. Πρόεδρος, ευχαριστούμε αγαπητοί συνάδελφοι και τώρα περνάμε στο επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη που είναι το σημείο 4. Είναι μια έκθεση πρωτοβουλίας σε σχέση με τις πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις στην Ουγγαρία. Ο κύριος Ρούι Ταβάρης είναι ο εισηγητής. Όπως γνωρίζετε, στις 16 Φεβρουαρίου η Ολομέλεια ε, ενέκρινε ψήφισμα με το οποίο ζητούσε από τη δικιά μας την Επιτροπή να παρακολουθήσει τα σοβαρά θέματα τα οποία αναφέρει το ψήφισμα αυτό και αφού ερευνήσει την κατάσταση να ετοιμάσει έκθεση με τα συμπεράσματά της. Σήμερα έχουμε την πρώτη ανταλλαγή απόψεων για το θέμα αυτό. Θα επικεντρωθούμε στην μέθοδο εργασίας που θα ακολουθήσουμε. Κύριε Τάβαρος, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Όπως αναφέρατε κι εσείς, αυτή είναι η πρώτη ανταλλαγή απόψεων που έχουμε για την έκθεση αυτή όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον πλουραλισμό ή όπως ε, τα αναφέρει το ψήφισμα της 16ης Φεβρουαρίου. Πρόκειται για τις αξίες, για την άσκηση της δημοκρατίας και το κράτος δικαίου στην Ουγγαρία. Σήμερα θα μιλήσουμε για την μεθοδολογία που θα ακολουθήσουμε. Ως εισηγητής, να ξέρετε ότι θέλω να ακούσω τις απόψεις των πολιτικών ομάδων όσον αφορά την μέθοδο εργασίας που θα ακολουθήσουμε, τη μεθοδολογία μας δηλαδή. Βλέπετε η έκθεση αυτή έχει κάποιες ιδιαιτερότητες, ιδιαιτερότητες που όλοι γνωρίζουν. Θα σας πω πώς βλέπω εγώ τη στάση που θα έπρεπε να κρατήσω ως εισηγητής. Αρχίζω με τρεις γενικές παρατηρήσεις. Πρώτον, βλέπω την έκθεση αυτή αμερόληπτα. Δηλαδή πιστεύω ότι η έκθεση αυτή δεν πρέπει να είναι μια έκθεση δεξιά από τη μία αριστερά από την άλλη, δεν είναι θέμα ιδεολογικό, είναι θέμα κοινών αξιών που επιτρέπουν σε όλους μας να συνεπάρχουμε εδώ, είτε είμαστε από τη δεξιά είτε από την αριστερά. Οπότε αυτό είναι το πρώτο μου σημείο. Αμεροληψία όσον αφορά την έκθεση αυτή. Η δουλειά λοιπόν πρέπει να βασιστεί στις κοινέ μας αξίες. Δεύτερη παρατήρηση. Πρέπει να βασιστούμε σε γεγονότα, νομικά, πολιτικά, Άρα αυτό θα είναι και το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα λειτουργήσουμε. Η Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, η συνθήκη της Λισαβόνας και βέβαια η δικιά μας προβληματική μέσα στο Κοινοβούλιο για το πώς βλέπουμε τα πράγματα μετά από τη θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας. Τρίτο θέμα. Τι στάση πρέπει να κρατήσουμε εμείς απέναντι στην έκθεση αυτή. Θα πρέπει να είναι σεβασμός και συνεργασία, διαφάνεια και συνεργασία με την Ουγγρική κυβέρνηση και την Ουγγρική κοινωνία των πολιτών, αλλά και με το Συμβούλιο της Ευρώπης, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και βέβαια και μέσα στο Κοινοβούλιο πρέπει να συνεργαστούμε με όλες τις κοινοβουλευτικές επιτροπές, πολιτιστική, δικαιοσύνη κλπ. Τέλος και μέσα σε αυτήν εδώ την Κοινοβουλευτική Επιτροπή εννοείται ότι πρέπει να συνεργαστούμε πλήρως ε, μεταξύ μας όλες οι πολιτικές ομάδες. Όπως όμως είπα και στην αρχή, θέλω να ακούσω τώρα και τη γνώμη των συναδέλφων. Τι ιδέες έχουν εκείνοι και πώς βλέπουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο θέλουν να λειτουργήσουμε προετοιμάσοντας την έκθεση αυτή. Η έκθεση αυτή έχει να κάνει με πολύ σοβαρά θέματα και γι' αυτό και πρέπει ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να την πάρει πάρα πολύ στα σοβαρά είναι θεμελιώδη δικαιώματα, δημοκρατία, κράτος δικαίου, που δεν έχουν να κάνουν μόνο με την Ουγγαρία, αλλά και με ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είναι μια τεράστια ευθύνη για μας να έχουμε αναλάβει την έκθεση αυτή. Μια ευθύνη που οι πολίτες θέλουν να την αναλάβουμε και να τη φέρουμε σε πέρας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτά λοιπόν εισαγωγικά και παρακαλώ τις πολιτικές ομάδες να μου πούνε τη γνώμη τους. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κύριε Ταβάρης. Έχω τρεις στον κατάλογο μιλητών. Φαγιό, Σβέμπερ και Βαρόν. Πρώτα η κυρία Φαγιό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Ρουή, για αυτά που είπες. Θα σας παρουσιάσω τη θέση του Χουάν Φερνάντο Λόπες Αγγιλάρ, που είναι ο σκιώδης εισηγητής της ε, ομάδας μας, αλλά που δυστυχώ δεν μπορεί να είναι εδώ σήμερα γιατί είχε ανηλυμένε υποχρεώσει. Θα προσπαθήσω όμω να σα παρουσιάσω τις δικές του απόψει που έχουμε συζητήσει μαζί. Είναι πολύ καλό που μπορούμε να αρχίσουμε την εκπόνηση της έκθεσης αυτής και πρέπει να γνωρίζουμε ότι το αντικείμενο της έκθεσης αυτής συνάδει απόλυτα με τις αρμοδιότητές μας. Όντως, εμείς ε, μπορούμε να προσφέρουμε πολύ σημαντικό έργο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θέλουμε ιδιαίτερα να υπογραμμίσουμε ότι στόχος μας δεν είναι να κρίνουμε μια χώρα και μια κυβέρνηση, αλλά να αναλύσουμε κατά πόσο οι τελευταίες δεχματικές μεταρρυθμίσεις στην Ουγγαρία είναι συμβατές με τις αρχές που αναφέρονται στη συνθήκη της Λισαβόνας και στη Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Δηλαδή, πρόκειται εδώ πέρα για το θέμα του πιο δίκαιο υπερτερή, που είναι το ευρωπαϊκό δίκαιο. Οτιδήποτε άλλο σκεφτεί κανείς θα ήταν αρνητικό και θα έχει αρνητικό αντίκτυπο ε, στους κατοίκους της ε, Ουγγαρίας. Θέλω να αναφερθώ και εγώ στα αρθρεπτά που μιλάει για το έργο της Επιτροπής και του εισηγητή. Εμείς πιστεύουμε και στόχος μας δεν είναι να τιμωρήσουμε μια χώρα μέλος, αλλά να κρίνουμε κατά πόσο υπάρχει ενδυνάμει κίνδυνος απέναντι στην ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις αξίες. Και γι' αυτό η προσέγγισή μας στη διαδικασία που ξεκινάμε τώρα να είναι ουδέτερη, να μην προκαταλαμβάνουμε το τι θα κάνουμε. Και εδώ δεν πρόκειται μόνο για το άρθρο 7. Το άρθρο 7 είναι ένα εργαλείο που έχουμε στη διάθεσή μας, δεν θα έπρεπε όμως να μονοπολίσει την έκθεση αυτή. Ο συγητής μας λέει ότι θέλει και ειδικέ ακροάσεις για να ασχοληθούμε με τα διάφορα θέματα που μας απασχολούν. Ναι, και εγώ θα έλεγα να οργανώσουμε και ένα ταξίδι στην Ουγγαρία που θα μας βοηθούσε να δούμε από πιο κοντά την πραγματικότητα της χώρας. Όσον αφορά την ουσία, ο εισηγητής έθεσε το θέμα της ανεξαρτησίας της δικαστικής αρχής μετά από τις συνταγματικέ μεταρρυθμίσεις και τις αρμοδιότητες που έχει αυτή η δικαστική εξουσία. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει ανεξαρτησία η οποία μπορεί να επιτευχθεί με τις κατάλληλες νομικές αλλαγές. Έτσι, όμως όπως έχει το σύστημα σήμερα, δεν φαίνεται αυτό, μια που ορίζεται ο δικαστής ε, από πριν. Η ανεξαρτησία της δικαστικής αρχής όντως θα πρέπει να είναι στην καρδιά της έκθεσής μας και να φαίνεται ότι είμαστε υπέρ της διάκρισης των εξουσιών που είναι βασικός πυλώνας της δημοκρατίας. Ένα άλλο θέμα είναι ο πλουραλισμός στα μέσα ενημέρωσης. Σε διάφορες εκθέσεις μας εμείς έχουμε πει ότι δεν πρέπει να υπάρχει ανάμειξη στα μέσα ενημέρωσης. Γιατί είναι βασικό στοιχείο αυτό για τη δημοκρατία. Το έχουμε πει ξανά και έχουμε συζητήσει ξανά και ξανά για τον νόμο που αφορά τα μέσα ενημέρωση στην Ουγγαρία. Η έκθεση αυτή λοιπόν πρέπει να ασχοληθεί και με το θέμα αυτό της ελεύθερης έκφρασης και των μέσων ενημέρωσης στην Ουγγαρία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Βέμπερ, είναι η επόμενη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι έχουμε να κάνουμε με μία πραγματικότητα, είτε πρόκειται για χώρα, για ένα νομοθετικό κείμενο. Είναι κάτι με το οποίο πρέπει να συμβιώσουμε. Είμαστε υποκειμενικοί από τη φύση μας, άρα όταν αποτιμούμε τα πράγματα τότε λαμβάνουμε υπόψη την ε, συνολική μας πείρα. Δεν πρέπει να προδικάσουμε, να προδικάζουμε όμως τα πράγματα. Αυτό είναι ύψης της σημασίας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τη, τον εισηγητή για την εισήγηση. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή με αυτή την έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας Υπάρχουν πολλά σημεία που καλύπτονται από άλλους φορείς και θα πρέπει να έχουμε μία διευρυμένη άποψη για την κατάσταση στην Ουγγαρία. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη όλες αυτές τις εκθέσεις και εισηγήσεις από ανεξάρτητους οργανισμούς. Υποστήριξα την ιδέα της συνέχειας γιατί και σε αυτή την Επιτροπή έχουμε μία σειρά συζητήσεων και θα πρέπει να συνεχιστούν. Αν θυμάμαι καλά, συμφωνήσαμε ότι μελλοντικά σε μία συνάντηση της ΛΥΠΕ θα καλέσουμε και τον ε, πρώην ε, είπα το εκπρόσωπο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κάποιον από την ε, Επιτροπή της Βενετίας και όλους τους ηθήνοντες που μπορούν να μιλήσουν για συνταγματικά θέματα στην Ουγγαρία. Η Επιτροπή της Βενετίας επίσης έχει φτάσει σε ορισμένα συμπεράσματα. Θα πρέπει να συνεχίσουμε σε αυτή μας την πορεία. Επίσης να έχουμε πιο διεξοδικές συναντήσεις με εκπροσώπους από την κοινωνία των πολιτών και των ΜΜΕ στην Ουγγαρία, να ακούσουμε όλα τα συμβαλόμενα μέρη και να δούμε ποια είναι η γενικότερη σκέψη συλλογιστική ως προς την κατάσταση στην Ουγγαρία. Δεν μιλάμε για κυρώσεις, δεν μιλάμε για διδάγματα, αλλά θα πρέπει να δώσουμε μάχη για τις δικές μας αρχές και αξίες τη στιγμή που θεωρούμε ότι στη μία ή στην άλλη χώρα υπάρχει παραβίαση δικαιωμάτων. Γι' αυτό ο Σκιώδης θα συνεργαστούμε μεταξύ μας και με τον εισηγητή. Η κυρία Μορβάη. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, πιστεύω ότι πριν μπούμε στην ουσία αυτής της έκθεσης, δηλαδή τα ε, κομμάτια, συγκεκριμένα κομμάτια της Ουγγρικής νομοθεσίας, θα πρέπει να δούμε ζήτημα αρχής, κατά πόσο δηλαδή ε, θα λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι απαρτιζόμαστε από 27 κράτη-μέλη και μόνο στην Ουγγαρία το νομικό σύστημα ελέγχεται διεξοδικά από το Συμβούλιο της Ευρώπης και φορείς, ευρωπαϊκούς φορείς. Ποιος είναι ο λόγος. Πολλοί είπαν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να, είναι, να σέβεται τις δικές της αρχές. Μία από τις βασικές αρχές είναι η μη διάκριση, η έλλειψη διακρίσεων. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει διαφορά μεταχείρισης χωρίς αιτιολόγηση. Διάφοροι οργανισμοί, ευρωπαϊκοί οργανισμοί, έχουν πολύ αυστηρά κατόφλια και μετρήσεις για να ορίσουν τη, μια σαφή αιτιολόγηση. Πού έγκυται η δικαιολογία, η αιτιολόγηση αυτής της ε, διαφορετικής μεταχείρισης. Λοιπόν, είτε θα μπορέσετε να την αιτιολογήσετε, είτε αυτή η έκθεση δεν θα πρέπει να συνταχθεί. Δεύτερο, ένα άλλο θέμα ε, διάκρισης είναι ποια σημεία επιλέγεται της Ουγγρικής νομοθεσίας. Εγώ έχω ορισμένε ε, υποδείξεις. Υπάρχει ο νόμος της εγγύου ιδιοκτησίας στην ε, Ουγγαρία, ως προς τα αγροτεμάχια δηλαδή. Θα μπορεί κανείς να αγοράσει αγροτεμάχια από όπου και να προέρχεται Άρα θα υπάρξει ένα είδος επικισμού των αγροτεμαχίων μας. Δεν θα έπρεπε λοιπόν όλοι οι ευφυείς αυτοί οι θύνοντες να δώσουν πληροφορίες στην Ουγγαρία για το πώς να αποφύγει κάτι τέτοιο. Πρόκειται για χιλιοϊπωμένα ζητήματα. Είναι η πρώτη, είναι η δεύτερη φορά που εισβάλλουν οι θύνοντες στη χώρα μας ε, αποφαινόμενοι για το νομικό μας σύστημα. Το πρώτο έγινε μετά την αποτυχία του κομμουνισμού και δεύτερη φορά είναι παρούσα. Άκρος ενδιαφέρον. Δηλαδή, σας ενδιαφέρει να δείτε κατά πόσο αυτό το νομικό σύστημα δεν πλήττει. Πριν δεν έπλητε το κομμουνιστικό καθεστώς, υπήρχε ατιμορρησία, υπήρχε πλούτος. Οι πρώην ιδιοκτήτες δεν μπορούσαν να ανακτήσουν την ιδιοκτησία τους, ενώ οι κομμουνιστές μπορούσαν να ιδιωτικοποιήσουν γη και ακίνητα όπως ήθελαν. Τώρα έχουμε μια κυβέρνηση η οποία θέλει να προβεί σε θεμελιώδεις αλλαγές. Όχι αρκετές, άρα το προσπαθεί. Τώρα έχουμε ένα νέο κύμα εμπειρογνωμόνων και νομικών ηθινόντων. Ε, επειδή ασχολούμαι με τα δικαιώματα των γυναικών, ο συνήγορος Βλέπω ότι υπάρχει συναισθηματική κατάχρηση ή τρομοκρατία. Όταν ε, επισυμβαίνει κάτι τέτοιο, τότε ο θήτης δεν ικανοποιείται με το οτιδήποτε. Στην αρχή, ας πούμε, το θύμα θα πει «Μα εγώ μαγείρευα πέντε μέσα τη βδομάδα, καθάριζα το σπίτι, προσπαθεί να αιτιολογήσει τη θέση του το θύμα, αλλά το καλύτερο που θα είχε να κάνει το θύμα είναι να μην δίνει καθόλου επεξηγήσεις και να λέει θέλω ίση, ισόνομη θέση είμαι ισόνομος εταίρος και θέλω ίση μεταχείριση. Και τότε θα πρέπει, διαφορετικά, θα πρέπει κανείς να διαχωρίσει τη θέση του. Αυτό θέλω να κάνει και η κυβέρνησή μου, να πει αρνούμε κάθε συνεργασία και αν δεν συμφωνείτε θα αποχωρήσω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Έγγελ. Λοιπόν, ε, θα προσπαθήσω μετά από την ε, ρήξη να συμφιλιώσω τους εταίρους και γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την πολύ επικοδομητική προσέγγιση του και με την έκθεση αυτή και με άλλα θέματα των συναδέλφων πρέπει να πω ότι συμφωνώ διότι αυτή η έκθεση πρέπει να ε, είναι υπερκομματική. Ακόμη και αν ε, δόθηκε κάποια πολιτική χρειά στη συζήτηση, ε, ιδίω στις πρώτες φάσεις, ότι είναι μια αντιπαράθεση μεταξύ δεξιάς και αριστεράς, ενώ εμείς θέλουμε να αξιολογήσουμε αν ε, οι νομικές αρχές που σεβόμαστε όλοι εφαρμόζονται στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αλλά όπως είπε και η κυρία Βέμπερ προηγουμένως, βάσει όλων των στοιχείων τα οποία έχουν αξιολογηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από τις επιτροπές που εξέτασαν τα θέματα αυτά σχετικά με την Ουγγαρία και το κράτος της ε, που αναφέρονται εις το Σύνταγμα, εις τους θεμελιώδεις κανόνες, ή ε, τις θεσμικές ρυθμίσεις που απορρέουν από το Σύνταγμα και όπως είπε και ο εισηγητής, σε πνεύμα δικαιοσύνης ε, και ε, ανοίγματο ε, θα πρέπει να πούμε ότι ακόμη και αν έχουμε διαφορές με την ε, ερμηνεία ορισμένων θεμάτων δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει ότι η Ουγγρική κυβέρνηση έχει προθυμοποιηθεί να κοιτάξει τα επίμαχα θέματα και να τα ευθυγραμμίσει με την κοινοτική γραμμή και θα πρέπει στη συνέχεια να κάνουμε μία πλήρη και εκτενή έκθεση που να καλύψει όλα τα θέματα διότι εγώ πιστεύω ότι δεν είμαι ο μόνος που εκφράζει την άποψη αυτή. Δεν θα μου άρεσε εάν έπρεπε σε έξι μήνες ή σε ένα χρόνο ή σε ένα μισή χρόνο να επαναφέρουμε το θέμα. Πρέπει να λύσουμε το θέμα τελεσίδικα τώρα όσο πιο εκτενώς γίνεται και όσο πιο γρήγορα γίνεται. Δεν είναι όμως μία έκθεση του άρθρου 7. Είναι μία έκθεση η οποία προσπαθεί να αξιολογήσει αν οι παραπομπές στο άρθρο 7 είναι αιτιολογημένες ή όχι και όχι το αντίστροφο. Οπότε Ουσιαστικά εδώ ανταποκρινόμαστε στην έκκληση της Ολομελίας που ζήτησε από την Επιτροπή μας να εξετάσει εάν είναι σωστό να σκεφτόμαστε ή όχι ότι χρειάζεται μία διαδικασία του άρθρου 7. Επίσης πέραν αυτού δεν είμαι πολύ ένθερμος υποστηρικτής των ακροάσεων. Ήδη κάναμε δύο. Δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε πολλές ακόμη. Ε, και ε, μας έχουν πει τα βασικά στοιχεία και είδαμε ποιες είναι οι αντιφατικές απόψεις, άρα δεν, δεν ακούσαμε κάτι το πρωτοφανές. Επίσης είμαι αντίθετο στην ιδέα ενός ταξιδιού στην ε, Ουγγαρία ε, και ε, για, διότι όπως και με την εκμάθηση γλωσσών ίσως ε, θα εμπνευστούμε εάν εμποτιστούμε στον ουγγρικό πολιτισμό. Και με αυτό καταλήγω και θέλω να πω ότι είμαι έτοιμος να συνεργαστώ με τον εισηγητή βάσει αυτών των αρχών. Ευχαριστώ η κυρία Ιντφελτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν, θα ήθελα να σας ε, επαναλάβω αυτό που έχω πει πολλές φορές, ότι εδώ δεν συζητάμε την Ουγγαρία, αλλά τα βασικά δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως που είναι εγγεγραμμένα εις ε, συνθήκες και ζητούμε να εφαρμοστούν. Μοιάζει με τη συζήτηση που έγινε δύο χρόνια, εδώ και δύο χρόνια για την Ευρωζώνη. Δεν μας βασολεί η Ελλάδα, μας ενδιαφέρει το Σύμφωνο Σταθερότητος και όπως η κυρία Μορβάη που λέγουν ναι αλλά εδώ τα βάζετε με την Ουγγαρία θα σας έλεγα να ελέγξετε την ιστοσελίδα μου και θα δείτε ότι λέω ότι είναι ελάχιστες χώρες από τις οποίες δεν έχω κάνει ε, κοινοβουλευτικές ερωτήσεις για τη διάκριση των ομοφιλοφίλων ή ε, για ε, τα μέσα ενημέρωσης. Έχουμε κάνει ήδη ερώτημα στην Ιταλία σχετικά με το θέμα αυτό στην κυβέρνηση Μπολουσκόνη το 2000 Οπότε ε, υιοθετώ το, υιοθέτησα και το ψήφισμα εναντίον της χώρας μου τον προηγούμενο μήνα. Είναι θέματα αρχής. Εάν εμείς δεν κατακρίνουμε πρώτοι τον εαυτό μας δεν θα μπορέσουμε ποτέ να προοδεύσουμε. Εάν υπάρχουν ε, παραβιάσεις ε, των ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων από διάφορες κυβερνήσεις πρέπει να κοινόμαστε. Αλλά ένα θέμα που δεν έχει εξεταστεί στο παρελθόν δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να το συζητήσουμε σήμερα. Συμφωνώ με την κυρία Φαγιόν και τον κύριο Έγγελ ότι ουσιαστικά ο στόχος δεν είναι να εκινήσουμε τη διαδικασία του άρθρου 7 και νομίζω ότι ήδη μπορούμε να καταλήξουμε ότι Υπάρχει μία έλλειψη ε, παρκών εργαλείων στα κράτη-μέλη. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα, όχι. Δηλαδή, είτε υπάρχουν γενικά εργαλεία ή έχουμε το άρθρο 7. Οπότε πρέπει να βρούμε τρόπο να έχουμε περισσότερα νομοθετικά μέσα και ο εισηγητής έχει δίκιο που βασίζεται στα γεγονότα. Συμφωνώ με ό,τι είπε ο κύριος Έγγελ για την ε, πληθώρα των ακροάσεων. Έχουμε κάνει όντως πολλές ακροάσεις, πρέπει να σκουμποθούμε και να δουλέψουμε. Και το βασικό θέμα που θέλω να πω είναι ότι είναι μία δοκιμασία για την Ευρώπη διότι εδώ και δεκαετίες η Ευρώπη εφαρμόζει μάλλον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφαρμόζει μια σειρά πολιτικών. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα γινόταν συζήτηση αυτή ε, για το ε, αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κράτη-μέλη που δεν έχουν ε, συμμορφωθεί εις ε, τους κανόνες χρηματοδοτήσεως. Αυτό είναι κάτι το οποίο κάνει καθημερινά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα και εμείς πρέπει να σκεφτούμε τι μας απασχολούσε όταν καταρτήσαμε το έγγραφο σχετικά με το θέμα αυτό και πώς μπορούμε να το προχωρήσουμε. Η κυρία Μάκεντάι. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή για την προσέγγιση του και για το ότι ήθελε πρώτα να συζητήσουμε εδώ, να ξέρουμε όλη την μεθοδολογία του, την οποία και υποστηρίζω σε ένα μεγάλο βαθμό. Είναι σημαντικό να παραμείνουμε ήρεμοι, να μην αφήσουμε τη φόρτισή μας να κυριαρχήσει. Φαίνεται ισορροπημένη η προσήγηση του εισηγητή. Την προηγούμενη εβδομάδα, όταν συζητήσαμε για τα μέσα ενημέρωσης, ήταν πολύ σημαντικό αυτό που είπαμε, ότι δηλαδή πρέπει να αντιμετωπίζουμε όλες τις χώρες ε, στην ίδια βάση και να μην κάνουμε διακρίσεις επειδή πρόκειται για την Ουγγαρία. Να έχουμε την ίδια προσέγγιση για όλες τις χώρες. Τώρα όντως η συγγήτρια από την ομάδα του ECR θέλω να σας πω ότι πιστεύουμε πως είναι πολύ σημαντικό το τι κάνουν τα κράτη-μέλη και πιστεύουμε στην κυριαρχία τους. Όμως, όπως και οι υπόλοιποι στη διεθνή κοινότητα, έτσι και εμείς εκφράζουμε κάποιες ανησυχίες για τόσα συμβαίνουν στην Ουγγαρία και θέλουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να φέρει σε πέρα στις αρμοδιότητές της που είναι ένα θεματοφύλακα των συνδικών. Συνεπώς, πρώτον, εκείνοι να ολοκληρώσουν το έργο τους. Και εμείς συνεχίζουμε να πιστεύουμε πως δεν είναι η κατάλληλη στιγμή εμείς να έχουμε έκθεση πρωτοβουλίας για αυτό το θέμα. Ότι θα είναι δηλαδή καλύτερο να περιμένουμε πρώτα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει ολοκληρώσει το δικό της το έργο και μετά να δούμε. Πάντως, έχοντας ακούσει τον κόσμο στην Ουγγαρία, τελικά ε, θα συμφωνήσω με τους συναδέλφους που λένε ότι φτάνουν πια οι ακρόασεις, δεν χρειαζόμαστε άλλη μια ακρόαση. Αλλά Πρέπει να δείξουμε ότι λαμβάνουμε υπόψη μας ε, την ειδική συγκυρία που υπάρχει στη χώρα και ίσως γι' αυτό θα ήταν θετικό να πάμε στην Ουγγαρία και να δούμε από πρώτο χέρι το τι γίνεται και να μην βασιστούμε μόνο στα όσα φτάνουν στα αυτιά μας από εκεί. Εγώ συμφωνώ με εκθέσεις που έχουν να κάνουν με ολόκληρο το ευρωπαϊκό φάσμα και όχι που καταδεικνύουν το πρόβλημα σε μία συγκεκριμένη χώρα, για παράδειγμα για τα μέσα ενημέρωσης. Όπως και να έχει το πράγμα πάντως, θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να συνεργαστούμε με τους σκιώδες εισηγητέ και με τον εισηγητή, προκειμένου να καταλήξουμε σε μια καλή έκθεση. Η κυρία Ευχαριστώ. Νομίζω ότι πρέπει να εκφραστεί κανείς σαφώς για να αποφευθούν ε, παρανοήσεις. Και εδώ δεν πρόκειται μόνο για το θέμα της Ουγγαρίας, πρέπει όμως να, να αναρωτηθούμε και πάλι. Τα τελευταία 20 χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκπονήσει ορισμένες αξίες που, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παίζει μεγάλη σημασία, έχει επιτυχίες, όχι μόνο συμβολικά, είναι ένας ε, θεσμός μεγάλης αξίας και πρέπει να δούμε ε, πώς θα κινηθούμε υπάρχει ένα κράτος μέλος το οποίο παραβαίνει τις αρχές μας, άρα τι μελιγενέστε. Και νομίζω ότι αυτό δεν είναι συγκεκριμένα θέμα για την Ουγγαρία. Αλλά υπάρχει ο κίνδυνος και βλέπουμε ότι στην Ουγγαρία υπάρχει κίνδυνος για την ένομο τάξη. Και αυτό δεν είναι κάτι το τεχνητό. Ε, θεωρώ ότι είναι πολύ σοβαρή, πρέπει να είμαστε πολύ σοβαροί με ένα τόσο ε, ιδιάζωνο πρόβλημα, αλλά εδώ εμπλέκεται και το ευρωπαϊκό δίκαιο και πρέπει να κινηθούμε και να κάνουμε μία ε, έκθεση κατά πρωτοβουλία και να εξασφαλίσουμε ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει σωστά τη δουλειά της αλλά πρέπει να πω ότι υπάρχουν θέματα τα οποία δεν έχουν αναφερθεί εδώ, διότι εγώ παραδείγματο χάρη είχα αντιταχθεί σαφέστατα στο ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με το Συμβούλιο αποφάσισαν ότι από το 2013 θα διαγραφούν από το Ταμείο Συνοχής ε, ε, πόροι για την Ουγγαρία διότι υπάρχει μία αρνητική εξέλιξη του ελίματος. Ε, εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει μία δοκιμαστική ρήτρα για μελλοντική πολιτική συνοχής και το απευχόμαστε. Κάτι τέτοιο δεν πρέπει να συμβεί ε, υπάρχουν όμως αυτοί οι οποίοι αντιτίθενται και πρέπει να αναφερθούν. Και εγώ είμαι αντίθετο στο άρθρο 7, στη διαδικασία του άρθρου 7, αλλά κάτι πρέπει να κινηθεί στην Ουγγαρία και πρέπει να πιέσουμε για να υπάρχει αυτή η εξέλιξη. Πρέπει όμως να δούμε εάν θέλουμε να συνομιλήσουμε με την Ουγγαρία, με ποιους θα, θα συναλλαχθούμε, με τους συντηρητικούς, με τους εκπαιδευτικούς, αλλά πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ να μην γίνει μια κίνηση η οποία θα στρέφεται κατά της Ουγγαρίας συγκεκριμένα. Θα ήθελα να πω ότι μέχρι τούδε δεν άκουσα, δεν υπάρχει και μεγάλη διαφωνία. Δεν άκουσα αντίθετες γνώμες. Δεν υπάρχει πλήρη συμφωνία, αλλά συμβατότης απόψεων. Βεβαίως δεν μπορούμε να ε, δούμε διεξοδικά το θέμα από πλευράς ε, modus operandi με μια απλή ανταλλαγή απόψεων. Δεν μπορούμε να αρχίσουμε με συμπεράσματα για το πώς ε, δηλαδή θα πρέπει να προχωρήσουμε. Νομίζω ακούσαμε τις ε, πολιτικές ομάδες, ε, τις πολιτικές ομάδες πολλοί μίλησαν για ακροάσεις, αρκετές είχαμε μέχρι τώρα και ίσως θα πρέπει να μεταβούμε στην ε, Ουγγαρία για να προωθήσουμε ένα διάλογο με τους Ούγγρους και την κοινωνία των πολιτών. Αυτό έχει σημασία και για τις δικές μας γνώσεις. Δεν προδικάζουμε Ούτε έχουμε προκαταλήψεις. Πολλές πολιτικές ομάδες, μερικές πολιτικές ομάδες μίλησαν για ακροάσεις, ότι είχαμε, αρχι... είχαμε ε, αρκετές ακροάσεις και ίσως θα πρέπει να εισακουστεί το Συμβούλιο της Ευρώπης και η Επιτροπή της Βενετίας. Και εν πάση περιπτώσει είμαι στη διάθεσή σας για ανταλλαγές απόψεων ε, όποιος θέλει να το συζητήσουμε και όποιος θέλει να συνεισφέρει για αυτό το σημαντικό ζήτημα. Η κυρία Φαζάν, όπως και πολλοί άλλοι, είπαν ότι δεν πρόκειται για μία δακτυλοδεικτούμενη χώρα, αφορά, αφορά ολόκληρη την Ευρώπη. Η κυρία Φαζόν και ο κύριος ε, Έγγελ μίλησαν για το άρθρο 7 και είπαν ότι ε, ναι μεν αναφέρεται το άρθρο 7 αλλά δεν πρόκειται για έκθεση δυνάμει του άρθρου 7. Δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε λοιπόν, αλλά ούτε έχουμε και αιμονές. Η εργασία μας, το έργο μας αφορά πολλά περισσότερα. Επίσης, υπάρχει ευρεία συνένεση για τα βασικότερα ζητήματα που θα μας απασχολήσουν στα πλαίσια του πλουραλισμού των συνταγματικών αλλαγών και του δικαιοδοτικού συστήματος. Και υπάρχουν ε, επικαλύψεις, μάλλον υπάρχει συμφωνία απόψεων. Όπως είπε και η κυρία Βέμπερ, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την υποκειμενικότητά μας, όμως δεν προδικάζουμε και δεχόμαστε τον πλουραλισμό. Πρόκειται για μια ομαδική εργασία και αυτό ακριβώς τονίσαμε, ότι αυτή η συλλογική εργασία θα προωθηθεί έτσι ώστε να υπάρχει συμβατότητα. Η κυρία Μόρβαη μίλησε για, τη, για διακρίσεις, για διαφορά μεταχείρισης χωρίς πλήρη αιτιολόγηση και συμφωνώ εν μέρη. Εάν αντιμετωπίζουμε προβλήματα σε άλλες ευρωπαϊκές ε, χώρες και εάν η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ κρατήσει παθητική στάση, τότε δεν επιτελούμε το έργο μας. Άρα Πρόκειται για θέμα ισότητας και ίσης αντιμετώπισης ως προς την αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα των κρατών. Βεβαίως, όπως αναφέρθηκε πολλές φορές, είχαμε πολλά ψηφίσματα όπου κατονομάσαμε χώρες και κυβερνήσεις, όπως για την Ολλανδία. Αναφερθήκαμε στον Πρωθυπουργό Ριτά. Και όπως είπε και η κυρία Ιντβελτ, είχαμε ψηφίσματα για τη Λιθουανία, την Ιταλία και όπως επέκρινε και τη δική της κυβέρνηση, όταν στην Πορτογαλία απολύθηκε ένας δημοσιογράφος, τότε τον κάλεσα εδώ για να δείτε τι συμβαίνει στη χώρα μου και θα ε, ήθελα όλοι να κάνουν το ίδιο, από όποια χώρα και να προέρχονται. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους, τη, τη, την κυρία Μάκεντά και την κυρία Έρνστ. Η κυρίως εργασία αρχίζει τώρα Πρόκειται για την απαρχή μιας σημαντικής αποστολής που πρέπει να επιτελέσουμε και μετά από το διάλογο αυτό ε, θα πρέπει να προωθήσουμε έναν ευρύτερο διάλογο, ξεκινώντας από εδώ και κινούμενοι προς ε, άλλα ευρωπαϊκά άλλους ευρωπαϊκούς φορείς, ε, κρατικές αρχές και κοινωνία των πολιτών. και θέματα που άπτονται αυτού του ζητήματος του πλουραλισμού, των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της δημοκρασίας και του, του κράτους δικαίου. Επόμενο θέμα Στη μερίσια διάταξη έχουμε αργήσει κατά 15 λεπτά. Στρεφόμαστε στο σημείο 5, δέσμευση και δι... δέσμευση των προϊόντων εγκλήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα έχουμε μια παρουσίαση από την Ευρωπαϊκή Επίτροπη και για να μπορέσουν οι δικαστικές αρχές να δημεύουν προϊόντα εγκλήματος, η Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή στις 12 Μαρτίου 2012 έχει προβάλει μία πρόταση οδηγίας για τη δέσμευση και δίμευση προϊόντων εγκλήματος που θα αντικαταστήσει το παρόν νομοθετικό πλαίσιο. Θα δώσω το λόγο λοιπόν σε εκπρόσωπο της Επιτροπής, τον κύριο Πρίμπε, ο οποίος θα μας ε, επεξηγήσει λεπτομερώς το περιεχόμενο και τον στόχο αυτής της πρότασης. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Πρίμπακ, θα ήθελα να ζητήσω από τους συναδέλφους που θέλουν να αποχωρήσουν να το κάνουν σύντομα, για να μπορέσουμε να εργαστούμε. Ο κύριος Τρίμπε έχει το λόγο και μετά θα συνεχίσουμε με διάλογο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω την Επιτροπή Λίμπε διότι υποστηρίζει τις προτάσεις της Επιτροπής για τη δίμευση και ανάκτηση προϊόντων, παρομοίων προϊόντων το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με βάση την δική του έκθεση, έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας για την αντιμετώπιση του εγκλήματος και το πρόγραμμα της Στοκχόλμης ζήτησε άμεση δράση για την αντιμετώπιση του θέματος. Διακόπτει ο Μιλών μέχρι να αποχωρήσουν οι υπόλοιποι. Thank you, sorry. Please. Με συγχωρείτε, σας ξαναδίνω το λόγο. Θα ξαναπροσπαθήσω, Πρόεδρε. Αναφέρθηκα στο γεγονός ότι η πρότασή μας ε, ε, ανταποκρίνεται στην έκκληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από την έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος και της πρότασης δυνάμει του προγράμματος της Στοκχόλμης και τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το 2010 για τη δίμευση προϊόντων εγκλήματος έτσι ώστε να ενισχύσουμε το νομικό πλαίσιο. Όπως ξέρετε, κάθε χρόνο υπάρχει παράνομος πλούτος, ο οποίος δημιουργείται, ο οποίος δεν μπορεί να αποτιμηθεί ποσοτικά και μόνο σε ορισμένα κράτη-μέλη έχουμε αριθμητικά στοιχεία. Στην Ιταλία το οργανωμένο έγκλημα έφτασε σε 150 δις ευρώ κέρδη το 2011 και στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2006 τα έσοδα ανέρχονταν σε 15 δις ε, λίρες τερλίνες. Επίσης γνωρίζουμε ότι ομάδες εγκλήματος δρούν διασυνοριακά σε άλλα κράτη-μέλη. Σύμφωνα με τα εκτιμώμενα εκτιμόμενα έσοδα, μπορούμε να κρίνουμε ότι το διμεθέν προϊόν είναι πολύ χαμηλό. Το 2006 στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε 125 εκατομμύρια τα οποία δημεύθησαν και κατασχέθηκαν τη στιγμή που μιλάμε για συνολικά έσοδα της τάξης του, των 15 δις. Το 2009 το διμευθέν προϊόν ανέρχεται σε 189 εκατομμύρια ευρώ και 195 αντιστοίχως Γαλλία και Αγγλία. Σήμερα βλέπουμε ότι τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας δεν επαρκούν για τη δίμευση και κατάσχεση προϊόντων εγκλήματος. Και γι' αυτό ανακύπτει και η ιδέα μιας νέας πρότασης. Τα περιουσιακά στοιχεία που δημεύονται είναι ανεπαρκή και η οδηγία δεν έχει εφαρμοστεί πλήρως. Έχει συσταλτική δε ερμηνεία σε πολλά κράτη-μέλη. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εγκρίθηκε στις 12 Μαρτίου για οδηγία για τη δίμευση και κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων εγκλήματος θα καταστήσει ευκολότερη τη δίμευση αυτών των περιουσιακών στοιχείων. Η οδηγία θέλει να δώσει οικονομικά κίνητρα για να προστατεύσουμε την, την ευρωπαϊκή οικονομία από την διείσδυση εγκληματικών στοιχείων και περιουσιακών στοιχείων αυτών. Επίσης, βασιζόμαστε στις ε, βέλτιστες πρακτικές και στις διεθνείς συμφωνίες για να καλύψουμε τα χάσματα με βάση τους υπόπτους και καταδικαστέντες. Επίσης, ορίζουμε καλύτερους ε, κανόνες για την επεκτεταμένη ε, δίμευση, δηλαδή δημεύσεις που δεν σχετίζονται με ένα και μοναδικό έγκλημα, αλλά απορρέουν από εγκληματικές δραστηριότητες ε, δυνάμει της δραστηριότητας των καταδικασθέντων. Επίσης, μιλάμε και για κατασχέσεις τρίτων μερών, έτσι ώστε να κατασχεθούν περιουσιακά στοιχεία, τα οποία μετέφερε ο ύποπτος σε κάποιον τρίτο. Έτσι, θα αντιμετωπίσουμε την ε, δραστηριότητα κατηγορουμένων ή υπόπτων που μεταφέρουν περιουσιακά στοιχεία σε συγγενικά πρόσωπα για να αποφύγουν τη δίμευση. Επίσης, σε περιορισμένες περιπτώσεις, όταν δεν υπάρχει καταδίκη, θα πρέπει να δημεύονται τα στοιχεία παρόλα αυτά. Και αυτό σε περίπτωση θανάτου ή επειδή κάποιος είναι φυγόδικος. Στη συνέχεια, οι αρμόδιες αρχές, ε, οι εισαγγελικές αρχές θα πρέπει να μπορούν να δημεύουν στοιχεία μετά από δικαστικές αποφάσεις. Η διαδικασία παγώματος θα προωθηθεί σε σοβαρές ε, υποθέσεις έτσι ώστε να μην μπορούν να διαφύγουν τα κεφάλαια της τελικής δήμευσης. Η οδηγία θα επιτρέψει στις αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές να συνεχίσουν τις έρευνες μετά από την εντολή δίμευσης, αλλά χωρίς να έχει εκτελεστεί πλήρως, διότι πολλές φορές αποκρύπτονται τα περιουσιακά στοιχεία και βγαίνουν στην επιφάνεια πολλά χρόνια μετά. Η οδηγία επίσης περιλαμβάνει διατάξεις για παγωμένα στοιχεία ενεργητικού έτσι ώστε να μην χάσουν την οικονομική τους αξία πριν δημευθούν ή κατασχεθούν. Και τέλος, η πρόταση θα εξασφαλίσει ώστε τα παγωμένα στοιχεία ενεργητικού να την κάνουν προστασίας μέσα στα πλαίσια του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Η, η πρόταση θα υποβληθεί στο Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων και Δικαιοσύνης τον Απρίλιο και ελπίζουμε, βασιζόμαστε στην υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις επερχόμενες διαπραγματεύσεις, έτσι ώστε και τα δύο θεσμικά όργανα να μπορέσουν να καταλήξουν σε αυτή τη νέα πρόταση. Ευχαριστούμε τον Τώρα, Θέλει κάποιος το λόγο, παρακαλώ. Δεν βλέπω. Συνεπώς, ευχαριστούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα όσα μας είπε και στη συνέχεια θα πρέπει να ορίσουμε εισηγητή. τώρα περνάμε στο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Αλλά εισηγητής φαίνεται ότι δεν είναι εδώ ακόμα. Συνεπώς, το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη, μετά από αυτό, ήταν για τις 5 μάλλον το προηγούμενο θέμα, για τις 5. Δεν είναι εδώ όμως. Είχαμε προβλέψει περισσότερο χρόνο για το σημείο 5 που δεν μας χρειάστηκε τελικά. Συνεπώς, προτείνω. Do we have... Do we... Do we have the legal uh, service here? Είναι εδώ η νομική υπηρεσία. Γιατί αν είναι εδώ η νομική υπηρεσία, ίσως θα μπορούσαμε να αλλάξουμε τη σειρά και να πάρουμε πρώτα το σημείο 7 και μετά το σημείο 6. Δεν είναι εδώ όμως η νομική υπηρεσία. Τότε λοιπόν θα πρέπει να διακόψουμε για λίγο μέχρι τις 5. Στις 5 θα συνεχίσουμε όταν θα είναι εδώ και ο εισηγητής μας. Okay, uh, now after this, uh, Καλώς, λέει η Πρόεδρος, μετά από αυτήν την σύντομη διακοπή μπορούμε να συνεχίσουμε. Ο εισηγητής, ο κύριος Μέλλο, μόλις ήρθε. Οπότε μπορούμε να εξετάσουμε το σημείο 6 στην ημερήσια διάταξη που είναι Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας σε υποθέσεις. Πρόκειται για μια οδηγία που βασίζεται σε μια πρωτοβουλία ορισμένων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πολύ σημαντικό θέμα όσον αφορά το ποινικό δίκαιο που θα καθορίσει τελικά πώς θα εφαρμόζεται η έννοια της αμοιβαίας αναγνώρισης όσον αφορά το ποινικό δίκαιο. Ο εισηγητής, ο κύριος ε, Μέλο, ορίστηκε για αυτό το θέμα και σήμερα θα έχουμε μαζί του μια ανταλλαγή απόψεων Έχουμε ήδη κάποιες τροπολογίες. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Μέλο πάντως πρώτα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ε, ζητώ συγγνώμη, αλλά έφτασα και λίγο νωρίτερα από την προτινόμενη ώρα. Βλέπω ότι και ο κύριος ε, Άλμπρεχτ ε, ήρθε νωρίτερα. Λείπουν ένα-δύο σκιώδεις. Τι θέλετε να περιμένουμε δύο-τρία λεπτά μέχρι ότου έρθουν και όλοι οι σκιώδεις στις 5 και 4 ή θέλετε να μιλήσω τώρα, να κάνω την εισήγησή μου τώρα και ενδεχομένως να επαναλάβω μενα στοιχεία. If Εάν προσέλθουν βέβαια και άλλοι σκιώδεις. Διαφορετικά ούτε καν δίλημα υπάρχει. Ωραία, ας αρχίσουμε τότε, ας Διαφορετικά θα καθυστερήσουμε πολύ. Θα μιλήσω στη μητρική μου γλώσσα, στα πορτογαλικά. Θα ήθελα να σας πω το εξής. Καταρχήν δεν θα ήθελα να επαναλάβω τα όσα προελέχθησαν στην ε, προηγούμενη συνεδρίαση για την οδηγία αυτή. Υπάρχουν νέα στοιχεία τα οποία θα μπορούσαμε να λάβουμε υπόψη και επ' αυτών θα ήθελα να αποφανθώ. Θα ήθελα καταρχήν να πω ότι δέκα βουλευτές υπέβαλαν τροπολογίες και εδώ συμπεριλαμβάνεται και ο υποφαινόμενος. Πρόκειται για στοιχεία πολύ επιμερισμένα. ως προς ε, ειδικέ πτυχές της οδηγίας. 54 ε, τροπολογίες έχουν υποβληθεί. Στο μεταξύ συναντηθήκαμε με τους σκιώδεις, με εκπροσώπους της Επιτροπής, του Συμβουλίου και της Προεδρίας. Αρκετές φορές συναντηθήκαμε. Είχαμε λοιπόν κοινέ συναντήσεις και από αυτές τις ε, συζητήσεις ανέκυψαν πολλά. Μπορώ λοιπόν να δεχτώ προσθήκες σε σχέση με τις ε, τέσσερις ε, τροπολογίες που έχω υποβάλει εγώ και σε σχέση με τέσσερα τμήματα αυτής της οδηγίας. Και θα ήθελα να σταθώ σε αυτά τα νέα στοιχεία, γιατί ως προς τα υπόλοιπα δεν έχετε παρά να αναγνώσετε το κείμενο. Το άρθρο υπαριθμών 5 γίνεται λόγος για την αναλογικότητα. Και ως προς την αναλογικότητα, θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει να αποτιμηθεί από τη χώρα έκδοσης και όχι από τη χώρα εκτέλεσης. Μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας και έχει σημασία που εκδίδεται αυτή η εντολή. Γι' αυτό θα πρέπει το κράτος έκδοσης να ενεργήσει εμπροκειμένο ως ανακριτική αρχή. Και γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να δούμε ποια είναι η διαφοροποίηση σε σχέση με το κράτος εκτέλεσης. Γι' αυτό το κράτος εκτέλεσης μπορεί να αποφανθεί σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε σχέση με το κράτος έκδοσης. Ως προς τη διπλή κατηγορία, σε σχέση με την διπλή κατηγορία. Εμείς όταν αποτιμούμε μία οδηγία ή οποιαδήποτε νομοθετικό κείμενο, θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και άλλα νομικά καθεστώτα, τα οποία θα μπορούσαν να είναι και ασύμβατα. Υπάρχει λοιπόν μία διαδικασία σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας. Μια πάγια διαδικασία. Επειδή πρόκειται για το ίδιο επίπεδο εφαρμογής, όταν μιλάμε για εγκλήματα είτε υπάρχει παράδοση φυσικών προσώπων και γι' αυτό ακριβώς μέσα στα πλαίσια της παράδοσης θα πρέπει να ισχύει το ίδιο νομικό καθεστώς δεν θα είχε νόημα να υπάρχει μία ε, ευρωπαϊκή εντολή έρευνας την οποία θα μπορούσε να αποτάξει ένα κράτος μέλος. Όταν λοιπόν πρόκειται για διπλή, διπλής τάξης κατηγορία, θα πρέπει να δούμε την εμβέλεια της Ευρωπαϊκής Εντολής Έρευνας. Γι' αυτό θα ήθελα να αναφερθώ στην τροπολογία μας. Δηλαδή ότι η Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας έχει καθολική αναγνώριση και στη χώρα ακρόασης μπορεί να τύχει άρνησης εάν στα πλαίσια της έρευνας γίνει λόγος για πλημελήματα που δεν αποτελούν έγκλημα στο κράτος εκτέλεσης. εκτός, και εδώ υπάρχει το μεγάλο εκτός, εκτός για την περίπτωση του 2-2. Δηλαδή, εκτός από το, τη συμφωνία του 2002 1584 της 13ης ε, Ιουνίου 2002 σε σχέση με τη διαδικασία έκδοσης μεταξύ κρατών μελών. Μιλάμε λοιπόν για 32 είδη εγκλημάτων που δεν υπόκεινται, υπόκεινται στον έλεγχο της διπλής κατηγορίας. Μιλάμε για έγκλημα όπως το οργανωμένο έγκλημα, το, την τρομοκρατία, την δουλεμπορία, την διακίνηση ναρκωτικών, την ε, ανθρωποκτονία εκ προμελέτης και ούτω καθεξής. Πρόκειται λοιπόν για εγκλήματα μεγάλης εμβέλειας, κοινωνικής εμβέλειας. Σε αυτή την περίπτωση ορίζεται ένα παράλληλο καθεστώς με αυτό της Ευρωπαϊκής Εντολής Έρευνας. Μία άλλη πολύ σημαντική τροπολογία έχει να κάνει με την κεντρική πτυχή της οδηγίας, διότι μιλάμε για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων και ελευθεριών και για εγγυήσεις που θα πρέπει να δοθούν στον υποδιερεύνηση και το δικαίωμα προσφυγής, δηλαδή ο υπόδικος θα μπορούσε να ζητήσει την εκτίμηση ενός δικαστηρίου για την δική του υπόθεση. Επειδή λοιπόν θέλουμε να είμαστε πολύ προσεκτικοί, θα θέλαμε να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα χρησιμοποιήσουμε μέσα παρακόλλησης για την εφαρμογή αυτής της οδηγίας, η οποία θέλει να είναι αποτελεσματική ως προς τη διερεύνηση του εγκλήματος και τη διασυνοριακή εγκληματικότητα στα κράτη-μέλη διότι δεν υπάρχουν σύνορα στο έγκλημα, ούτε περιορίζεται στο χώρο Σέγγεν. Η εγκληματικότητα είναι ρευστή, είναι ολοένα και πιο διασυνοριακή και γι' αυτό πολλές φορές η δικαιοσύνη χάνει μηχανισμούς αντιμετώπισης μέσα στα πλαίσια των δικαιοδοτικών συστημάτων. Γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία να εφαρμοστεί αυτή η οδηγία και τι θέλουμε να κάνουμε με τις ε, προσφυγές. Οι αντίδικοι να μπορούν να προσπίσουν τα δικαιώματά τους. Αυτό είναι το πρώτο σημείο. Επίσης, οι προσφυγές να μην είναι μέσον παρακόλλησης, το οποίο να καταπνίξει την οδηγία σαν τρίτο σημείο οι αντίδικοι να πρέπει πάντα να πληροφορούνται για τα δικαιώματά τους, δηλαδή οι υπόδικοι θα πρέπει να γνωρίζουν τι δικαιώματα έχουν πλήρως και θα πρέπει επίσης να εγγυηθούμε το απόρριτο της διερεύνησης ή το, της ανάκρισης από το κράτος έκδοσης. Έτσι ώστε να φτάσουμε σε αίσιο πέρας. Βασίζομαι λοιπόν στην πείρα μου Και θέλω ακριβώς να σταθμίσω όλα αυτά τα συμφέροντα, στα πω έτσι. Δηλαδή, θα πρέπει να δούμε κατά πόσο το δικαίωμα και το δίκαιο να μην είναι ανασταλτικού χαρακτήρα. Άρα θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα εκτέλεσης και τη στιγμή που γίνεται προσφυγή θα πρέπει να υπάρχει μία δυνατότητα, συγκεκριμένη δυνατότητα προσφυγής και γι' αυτό μιλάμε για μία ανασταλτικό χαρακτήρα και άρα εκτελείται η Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας, αλλά τα αποδεικτικά στοιχεία αποστέλλονται στην χώρα έκδοσης μετά από την τελική απόφαση. Γι' αυτό μιλάμε για έναν χρόνο, για ένα συγκεκριμένο χρόνο μέχρι να φτάσουμε σε μία απόφαση χωρίς να υπάρχει παρελκυστική τακτική. Πολλές φορές όμως από τη χώρα έκδοσης μπορούν να δημιουργηθούν βλάβες στον, στο υποέραυνα φυσικό πρόσωπο. Γι' αυτό θα πρέπει να γίνεται μία σωστή στάθμιση τη στιγμή που θεωρεί το φυσικό πρόσωπο υπό έρευνα ότι το μέτρο εκτέλεσης θα δημιουργήσει ανήκε στο βλάβη, μπορεί να ζητήσει αναστολή αλλά αυτό θα πρέπει να αποφασιστεί από μια δικαστική αρχή. Άρα δεν υπάρχει διαδικασία αναστολής, αλλά εάν ο ερευνόμενος, ο υποέρευνα θεωρεί ότι η υπέστη σοβαρή και αναπόδραστο βλάβη, μπορεί να ζητήσει την εφαρμογή της διαδικασίας αναστολής. Τέλος, το ίδιο μπορεί να υποθεί και, από ε, και για την πλευρά του κράτους έρευνας. Διότι η παρακράτηση των αποδεκτικών στοιχείων μπορεί να προδικάσει την ίδια την ε, έρευνα, να την επηρεάσει. Γι' αυτό, κατά τον ίδιο τρόπο που ο υπόδικος υποέρευνα μπορεί να ζητήσει απόφαση δικαστηρίου, το κράτος έκδοσης πρέπει να διαθέτει τα αποδεικτικά στοιχεία προς το κράτος εκτέλεσης. και να ζητηθούν αυτά τα αποδεικτικά στοιχεία πριν από την τελική απόφαση. και μίλησα για τις προσφυγές επί μακρόν, διότι είναι το κύριό μας μέλημα σε αυτή την οδηγία. Όταν η χώρα έκδοσης καταδεικνύει ότι ελοχεύει κίνδυνος κατά τη διάρκεια της διενέργειας της έρευνας, πριν από την τελική ε, απόφαση μπορεί να ζητήσει εγγύησεις έτσι ώστε στο τέλος της διαδικασίας, εάν ο υπόδικος κερδίσει τη δίκη, τότε τα, στοιχεία που, τα αποδεικτικά στοιχεία που απεστάλησαν είτε θα καταστραφούν, είτε θα επιστραφούν στο αρχικό κράτος, αλλά δεν θα μπορέσουν επουδενή να χρησιμοποιηθούν. Αυτό έτσι μάλλον διέπεται το καθεστώς προσφυγών και ως προς το, ε, τα δικαστικά έξοδα υπάρχει κόστος που βαρύνει τα κράτη. Και θεωρούμε ότι δεν θα ήταν σωστό το κράτος εκτέλεσης να πρέπει να επομιστεί όλα τα δικαστικά έξοδα με βάση την, ε, τις έρευνες που έχουν ήδη διενεργηθεί. Μιλάμε λοιπόν για το κράτος έκδοσης καταρχήν. Εάν λοιπόν το κράτος έκδοσης γνωρίζει ότι δεν καταβάλει, δεν συμμετέχει στα έξοδα, τότε η σχέση είναι ετεροβαρής. Και γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει επιμερισμός ανάληψης ε, εξόδων. Διαφορετικά το κράτος έκδοσης ε, δεν επομίζεται τίποτα. Επίσης, υπάρχουν ε, κράτη που αντιμετωπίζουν μεγάλα δημοσιονομικά προβλήματα και ελλείμματα και δεν μπορούν να αναλάβουν, να επομιστούν ένα τέτοιο κόστος. Γι' αυτό θα πρέπει να επιμεριστούν τα έξοδα και να τα αναλάβουν εξημισίας το κράτος έκδοσης και το κράτος εκτέλεσης. Και μπορούν τα κράτη, αν το συμφωνήσουν, να προβάλλουν ένα διαφορετικό καθεστώς. Ας πούμε, η Ιταλία με τη Μάλτα. Η Ιταλία έχει πολλές δυνατότητες έχει άλλο δημοσιονομικό εκτόπισμα σε σχέση με τη Μάλτα. Μπορεί λοιπόν να αναλάβει ένα μεγαλύτερο μέρος των εξόδων σε σχέση με τη Μάλτα. Και θα ήθελα τέλος να αναφερθώ σε κάτι που μας απασχολεί όλους. οι αρχές παρέμβασης θα πρέπει να είναι δικαστικές αρχές, δεν μπορεί να είναι αστυνομικές αρχές. Αυτός που αποφασίζει είναι μία δικαστική αρχή, ένα δικαστήριο, ένας δικαστής. Αυτό θα πρέπει να είναι απόλυτα σαφές. Το High Court of Justice του Ηνωμένου Βασιλείου της Δευτέρας Νοεμβρίου 2011 αποφάσισε ρητά και απερίφραστα υπέρ της αμοιβαίας αναγνώρισης και αμοιβαίας εμπιστοσύνης και έγινε λόγος για αποκλειστικά δικαστική αρχή η οποία μπορεί να αποφανθεί. Διαφορετικά δεν θα μπορούσε να εκτελεστεί μια ευρωπαϊκή εντολή έρευνας. Δεν μπορούμε να ενταχθούμε σε ένα διοικητικό, αλλά σε ένα δικαστικό πλαίσιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Mr. Mello. Ευχαριστώ. κύριε Μέλλο. Και τώρα πρώτα θα δώσω το λόγο στο Συμβούλιο στην κυρία Οκέν και μετά στην ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Το Συμβούλιο μελέτησε πολύ προσεκτικά τις ε, τροπολογίες και βλέπουμε ότι πολλές από αυτές ακολουθούν την προσέγγιση του Συμβουλίου και γι' αυτό θα αναφέρω τα πιο σημαντικά ε, για τα κράτη-μέλη. Ο κύριος Μέλο αναφέρθηκε στην αναλογικότητα και συμφωνούμε με τον κύριο Μέλο ότι θα πρέπει να γίνεται από τα εκδίδοντα κράτη, δηλαδή δεν πρέπει να επιτρέψουμε στο εκτελών κράτος να αξιολογήσει την αναλογικότητα σχετικά με το θέμα αυτό. Ε, υπάρχουν όμως άλλα μέτρα τα οποία χρειάζονται χέγγια για την εφαρμογή τους και η γενική προσέγγιση του Συμβουλίου είναι ότι πρέπει να εξετάσουμε το θέμα της αναλογικότητας πιο προσερμοσμένο κατά περίπτωση και με μέτρα τα οποία δεν θα είναι ε, πολύ επεμβατικά και εδώ αναφέρομαι στο άρθρο 3 και 4 του χάρτη των Γενικών Σχολείων του Συμβουλίου. Τα μέτρα αυτά μπορούν να αποτελέσουν βάση για περαιτέρω συζήτηση τόσο από πλευρά της αναλογικότητος και ως βάση για μία άρνηση και απόρριψη. Ένα άλλο βασικό θέμα για το Συμβούλιο που δεν αναφέρθηκε από τον εισηγητή είναι το θέμα της εμβέλειας της οδηγίας και θα πρέπει όλοι να γνωρίζουν ότι ο στόχος του Συμβουλίου είναι να έχουμε όσο δυνατόν περισσότερα μέτρα στο κείμενο κατά τρόπον ώστε να υπάρξει προστιθέμενη αξία στο ισχύον σύστημα. Ε, όσο αναφορά την ε, παρακολούθηση των τηλεπικοινωνιών. Αυτές είναι απαραίτητες για την καταπολέμηση ιδίως του, της, αυστηρή, της οργανωμένης εγκληματικότητας και θα πρέπει να περιληφθούν ή στην οδηγία και θα πρέπει συγχρόνως να σκεφτούμε ότι ακόμη και αν αποκλείσουμε ορισμένα μέτρα αυτό δεν σημαίνει ότι τα μέτρα αυτά δεν χρησιμοποιηθούν για να επιτύχει κανείς μία απόφαση από, τη, στα πλαίσια της οδηγίας θα αναφερθώ και σε άλλα θέματα τα οποία έθιξε ο κύριος Μέλο, δηλαδή για τα νομικά διορθωτικά μέτρα, τη δυνατότητα να διευκρινιστούν αυτές ε, οι νομικές ε, δυνατότητες επανορθώσεως που περιλαμβάνονται στην εθνική νομοθεσία αλλά θα πρέπει να ρυθμίζονται από το ε, ε, διεθνή νομοθεσία και οι μη δικαστικές ε, αρχές κατά τη γνώμη μας πρέπει να προχωρήσουν σύμφωνα με τη συμβιβαστική λύση την οποία επέτυχε το Συμβούλιο χωρίς να διακινδυνεύσουν την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης. Και η λύση αυτή την οποία έχουμε προωθήσει και ε, προχωρήσαμε στο Συμβούλιο θα επιτύχει και την ε, ευελιξία του μονίμου συστήματος. Τέλος θα ήθελα να τονίσω ότι η σύναψη αυτής της ε, οδηγίας ε, είναι πολύ σημαντική για το Συμβούλιο και με πολύ ενδιαφέρον θα συμμετάσχουμε σε περαιτέρω διαπραγματεύσεις για την ε, οδηγία αυτή. Ευχαριστώ. Εν ονόματι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τώρα ο κύριος Ολιβιέ Τέλ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή για τις εξηγήσεις αυτές που ήταν πολύ σαφείς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την θέληση του εισηγητή να ενισχύσει τα δικαιώματα των ατόμων και να προωθήσει ε, το σύστημα το οποίο να ακολουθεί τη σωστή κατεύθυνση ιδίως όσον αφορά την αναλογικότητα και την ε, έλλειψη ε, ελέγχου της διπλής εγκληματικότητος που προβλέπεται στις περιπτώσεις παραβάσεων ε, για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Πιστεύουμε ότι όλα αυτά ακολουθούν τη σωστή κατεύθυνση και είναι μια καλή ευκαιρία τώρα να σταματήσει αυτό το κατακαιρματισμένο σύστημα όσον αφορά τα ποινικά μέτρα και να ληφθούν οι υπόψη και τα σύγχρονα μέτρα τα οποία θα πρέπει να εξεταστούν από μια ευρωπαϊκή νομοθεσία για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τα θεμελιώδη δικαιώματα για την εκτέλεση ακριβώς και χρησιμοποίηση αυτών των συγχρόνων μέτρων που προτείνονται από τα κράτη-μέλη. Βεβαίως είμαστε στη διάθεση και του Συμβουλίου και ε, του Ευρωκοινοβουλίου σαν ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ε, προσφέρουμε βοήθεια και για τα μέτρα προστασίας των ατόμων και για την ολοκλήρωση των ερευνών και της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος. Ευχαριστώ. Και τώρα θα δώσω πρώτα το λόγο στον κύριο Άλμπρεχτ σαν ε, σκιώδη συγητή. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μέλο για την καλή συνεργασία Φαντάζομαι ότι ήδη έχουμε προχωρήσει διάφορα βήματα με αυτή την συνεργασία και ε, χρειάστηκε προσπάθεια για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο και ακόμη και αν συμφωνούμε σε διάφορα σημεία υπάρχουν άλλα τόσα τα οποία θα μας απασχολήσουν και στη συνέχεια και γι' αυτό απεδείχθη από τις τροπολογίες για το θέμα το οποίο μόλις τώρα έθιξε πάλι το Συμβούλιο, δηλαδή δηλαδή τις δυνατότητες στο κράτος εκτελέσεως να ελέξει την αναλογικότητα. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να συζητήσουμε και στη συνέχεια και θα επηρεάσει και τις διαπραγματεύσεις διότι είναι κάτι το οποίο θεωρούμε σαν απαραίτητο να υπάρχει δηλαδή έλεγχος της αναλογικότητας βάσει των μέτρων της της αμοιβαίας αναγνώρισης και από τη μία πλευρά είναι κάτι το οποίο πρέπει να εξεταστεί από πλευρά θεμελιωδών δικαιωμάτων και διαδικασιών αλλά και ιδίω βάσει της πείρας που έχουμε από το ένταλμα συλλήψεως ξέρουμε ότι συνθήκες όπου ε, ε, εμπλέκονται διάφορα νομικά συστήματα στη διαδικασία αυτή είναι κάτι το οποίο δεν γνωρίζουν ενδεχομένως τα άτομα τα οποία εμπλέκονται και γι' αυτό ε, το ε, ε, κράτος που εκδίδει την αίτηση, the issuing state αγγλικά, πρέπει ε, να συμμετάσχουν στη διαδικασία αλλά συγχρόνως ε, ε, οι εμπλεκόμενοι στο κράτος της εκτελέσεως θα πρέπει και αυτοί να συμμετάσχουν στη διαδικασία. Είναι κάτι που πρέπει να μας απασχολήσει ακόμη. Με αυτό είναι στενά συνδεδεμένο το θέμα των όρων της ε, απελάσεως που έχει διατυπωθεί όχι όμως επαρκώς ικανοποιητικά στην έκθεση και ερχόμαστε στη συνέχεια και στο πλαίσιο εφαρμογής αυτών των μέτρων, δηλαδή της ε, και καλυμμένης ε, ε, μεσολάβησης ε, το θέμα της ε, τηλεφωνικής παρακολούθησης δηλαδή πολλών ευαισθητών θεμάτων όπου πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί γιατί νομίζω ότι εδώ πρέπει να βελτιωθούν πολλά θέματα στα κοινά πρότυπα και στις κοινέ διαδικασίες για θέματα τα οποία πλήττουν τα θεμελιώδη δικαιώματα είναι κάτι που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και εφόσον έχουμε τη δυνατότητα να υπάρξει και μία νέα έκκληση προς το Συμβούλιο ώστε όσον αφορά το εκτελεστικό δίκαιο και τη συμμετοχή να τα τελειοποιήσει διότι μόνο όταν αυτά θα έχουν βελτιωθεί από το Συμβούλιο θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Ε, μία τέτοια αιρεσιμότητα δεν νομίζω ότι θα γίνει σε αυτό το στάδιο αποδεκτή από τους πολίτες κυρία Βέμπερ έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα μιλήσω εκ μέρους της κυρίας Σάρα Λάτφορτ που είναι η σκιώδης εισηγητριά μας. Ο καθορισμός μιας ε, περιοχή ενό χώρου δικαιοσύνη και προστασία των πολιτών μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι κάτι εύκολο, διότι υπάρχουν χώρες στις οποίες ισχύουν εντελώ διαφορετικές νομικές παραδόσεις και το να προσπαθούμε να τα συμβιβάσουμε αυτά δεν είναι τόσο εύκολο. Ακριβώς γι' αυτό και για να σας εξηγήσω ότι δεν έγινα σχιζοφρενής μέσα στις τελευταίες ώρες, πρέπει να σας πω ότι να, έχω δύο συναδέρφους οι οποίοι μου ζήτησαν να μιλήσω εκ μέρους τους αλλά οι δικέ τους οι θέσει είναι αντιφατικές μεταξύ τους ορισμένα σημεία. Σα το λέω για να καταλάβετε. Το έχω πει και σε αυτού, βέβαια. Αλλά ήθελα να σας ε, μεταφέρω τώρα τις απόψεις της τη γητριάς μα, της κυρίας Λάτφορντ, η οποία θεωρεί ότι σκοπός της Ευρωπαϊκής Εντολής Έρευνας είναι να καλύπτει όλα τα σχετικά μέτρα, αλλά να λαμβάνει υπόψη τις διάφορες ευαισθησίες. Κατά τη γνώμη της, οι έλεγχοι, οι μυστικές έρευνες δεν ανταποκρίνονται στον στόχο αυτό και γι' αυτό θέλει να αφαιρεθούν. Κατέθεσε διάφορες τροπολογίες προς αυτή την κατεύθυνση ίδια. Τώρα στην τροπολογία του αριθμού 24 ο εισηγητής εισαγάγει την ιδέα της αναλογικότητας. Η κυρία Λάτφορ το υποστηρίζει αυτό και στην τροπολογία της επί του άρθρου 5α προσθέτει και την ιδέα του μικρού παραπτώματος που μπορεί να διαφέρει από την αναλογικότητα. Θεωρεί ότι ένα μέτρο μπορεί να είναι δυσανάλογο. Ακόμα και αν δεν είναι μικρό το παράπτωμα, μπορεί να μην υπάρχει αναλογική αντιμετώπιση. Βέβαια, ο άλλος συνάδελφος διαφωνεί με αυτό. Όχι εγώ. Εδώ δεν σας παρουσιάζω τη δικιά μου άποψη καθόλου. Η κυρία Λάτφορ θέλει επίσης να υπογραμμίσουμε ότι τα μέτρα που έχουν να κάνουν ε, με τον αξιωματούχο της αστυνομίας δεν μπορεί να έχουν την ίδια σημασία ανάλογα με το σε ποια χώρα πάει. Συμφωνεί βέβαια με την ιδέα που λέει ότι είναι πολύ δύσκολο αυτό που αναφέρεται στο άρθρο 10 για την άρνηση. Συμφωνεί πάντως με τον εισηγητή για τη νέα απλοποιημένη δομή Όμως αν δεχτούμε την διπλή εγκληματικότητα είναι σαν να πηγαίνουμε πολύ μακριά τη δικαστική συνεργασία. Αυτή η διπλή εγκληματικότητα πρέπει να ελέγχεται εφόσον ε, τα μέτρα ε, το απαιτούν. Γι' αυτό και έχει υποβάλει σχετική τροπολογία προκειμένου να επιταχύνεται η συνεργασία μεταξύ διαφορετικών δικαστικών αρχών. Όσον αφορά τώρα την διόρθωση. Είναι σημαντικό τέτοια μέτρα να αναγνωρίζουν και να γίνεται η εκτέλεση σε περίπτωση που προβλέπει ο Εθνικός Νόμος την ενημέρωση πριν τεθούν σε εφαρμογή τα μέτρα. Και εδώ έχει μια τροπολογία, κύριε Λάτφορντ. Στην περίπτωση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης έχουμε δει μερικές φορές ότι δεν ακυρώνονται σωστά από τις δύο πλευρές ε, τα εντάλματα εφόσον έχει αποσυρθεί το θέμα. Ε, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί να μην συμβεί αυτό και στην περίπτωση της έρευνας. Για να υπάρχει νομική βεβαιότητα είναι σημαντικό η εντολή να ακυρώνεται και στη χώρα έκδοσης και στη χώρα εκτέλεσης έχει υποβάλει και διάφορες τροπολογίες για την προστασία δεδομένων και θεωρεί ότι είναι πολύ σημαντικό να αλλάξει την άποψή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να φροντίσει για την καλή μεταχείριση των προσωπικών δεδομένων. Για το θέμα της διόρθωσης τώρα, αν ένα άτομο δεν μπορεί να ενημερωθεί ενώ δικαιούται, τότε μειώνεται η αποτελεσματικότητα της διόρθωσης που του προσφέρεται. Και το τελευταίο που έχει να πει η κυρία Λάτφορντ είναι το εξή. Η πρακτική η οποία δεν χρησιμοποιείται πολύ στην Ευρωπαϊκή Αστυνομία, παρόλα αυτά πρέπει να υπάρχουν σαφείς κανόνες που να προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και εδώ λοιπόν έχει υποβάλει τροπολογίες προς αυτή την κατεύθυνση. Λέει επίση ότι είναι σημαντικό όταν ε, γίνεται μεταγωγή πρέπει να φροντίζουμε να μην είναι χειρότερες οι συνθήκες από ό,τι θα ήταν στη χώρα του. Τώρα έχω και τον κύριο Γιούτσετ εδώ, ο οποίος εκφράζει την ανησυχία του για το θέμα των μικρών παραβάσεων και για το άρθρο 10 που αναφέρεται στην βάση για άρνηση. Κατά τα άλλα, εύχομαι καλή τύχη στον κύριο Μέλο που θα προσπαθήσει να εικονοποιήσει όλους όσοι υπέβαλαν τροπολογίες. Ελπίζω να πετύχει ένα καλό σεβασμό. Ο κύριος Δεγιόν τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, λέει ο κύριος Δεγιόντ. Ευχαριστώ και εγώ τον εισηγητή, τον κύριο Μέλο. Και ζητώ συγγνώμη που κατέθεσα 40 τροπολογίες. Όντως είναι πολλές δεν το συνηθίζω. Δεν είναι όμως τόσο τρομακτικό όσο φαίνεται το πράγμα. Πρώτα απ' όλα, προσπάθησα να λάβω υπόψη μου τη γενική προσήγγιση που υπέβαλε το Συμβούλιο κάποια στιγμή. Δεν ξέρω αν η γενική προσέγγιση ήταν βελτίωση του αρχικού κειμένου. καλό είναι να διευκολύνουμε τις διαπραγματεύσεις που θα ακολουθήσουν. Πάντως υπάρχουν και ουσιαστικέ διαφορές. Τόσο η κυρία Βέμπερ ή τέλο πάντων οι μισές από την κυρία Βέμπερ αλλά και προλαλήσα το είπε ότι Στη χώρα μου, στις κάτω χώρες, το κοινοβούλιο είχε ζητήσει έρευνα γιατί τελικά η αστυνομία είχε καταλήξει να μην ξέρει τι κάνει με τις υποκλοπές και να έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που δεν θα έπρεπε μέσα στη δημοκρατία. Γι' αυτό τα μέτρα αυτά ελήφθησαν μετά από λεπτομερείς έρευνες και του Εθνικού Κοινοβουλίου. Προσοχή λοιπόν γιατί μπορεί να είναι επικίνδυνο να έχουμε μια ευρωπαϊκή προσέγγιση προς αυτή την κατεύθυνση στα πλαίσια της ε, ευρωπαϊκής ε, αυτής εντολής. Όταν έχουμε να κάνουμε με τις υποκλοπές και αν θέλουμε να μιλήσουμε για συμβιβασμό, το υλικό το οποίο ήδη είναι διαθέσιμο, δεν υποκλέπτεται δηλαδή, αλλά είναι αποδεικτικά στοιχεία τα οποία ήδη υπάρχουν, αλλά απορρέουν από υποκλοπές, θα μπορούσαμε ίσως να το δεχτούμε, αλλά όχι να γίνονται υποκλοπές με σκοπό να βρεθούν τα αποδεικτικά αυτά στοιχεία. Χρειάζεται έλεγχος αναλογικότητας και στις δύο πλευρές, λέει η κυρία Λάτφορτ, μα από την εμπειρία που έχουμε με το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψη μέχρι τώρα, δείχνει ότι υπάρχουν χώρες που το χρησιμοποιούν πάρα πολύ εύκολα. Υπάρχει στο σύστημα. Και πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ απογοητευτικό που παρά τη συζήτηση που έγινε στην Ολομέλεια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αλλάζει τίποτα στο τρέχον σύστημα και δεν φροντίζει να υπάρχουν περισσότερες εγγυήσεις ε, και στις δύο πλευρές, και στη χώρα έκδοσης και στη χώρα εκτέλεσης δηλαδή. Αυτό σημαίνει ότι τώρα θα έχουμε μία νέα πρόταση η οποία δεν μας δίνει εγγύησεις για αυτήν την ε, δοκιμασία αναλογικότητας. Πρέπει επίσης να σας πω ότι δεν έχει να κάνει μόνο με την αναλογικότητα, είναι και μια δοκιμή που γίνεται για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Και όταν μιλάμε για αμοιβαία εμπιστοσύνη, εφόσον αιτιολογείται τα ανθρώπινα δικαιώματα, νομίζω ότι είναι κάτι. Δεν μπορούμε απλώς να πούμε «Α, εμπιστεύομαι την άλλη πλευρά», γιατί έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα που τα πράγματα δεν πήγαν καλά. Υπάρχουν λοιπόν πολλά συγκεκριμένα ζητήματα, τα οποία είναι πολύ σημαντικά για τη δικιά μου ομάδα και κάποια άλλα πιο τεχνικά που έχω συμπεριλάβει στις τροπολογίες μου. Ο εισηγητής, δεν ξέρω, ας μου πει, νομίζω ότι αύριο θα είχαμε μια συνάντηση σχεδόν εισηγητών. Είναι έτσι? Εγώ πραγματικά πολύ θα ήθελα να έχουμε συζήτηση και συμβαστικέ τροπολογίε, Δεν ξέρω αν με ακούει όμω η συγητής. Έλεγα, κύριε Σιγητά, ότι θα ήθελα να έχουμε ανταλλαγή απόψεων μεταξύ μας για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Ευχαριστούμε κύριε Τεγιόνγκ και κυρία Χέιτ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σύμφωνα με την ε, πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι πολύ βασικό στα πλαίσια της διασωνοριακής εγκληματικότητας να υπάρχει συνεργασία για την καταπολέμηση ε, ιδίω όταν πρόκειται για εμπόριο ατόμων διότι υπάρχουν πολλοί τομείς στους οποίους χρειάζεται περισσότερη συνεργασία θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή διότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να συγκρίνει κανείς τα συστήματα των διαφόρων κρατών τα οποία είναι διαφορετικά και το θέμα της αμοιβαίας αναγνώρισης αποτελεί μια βασική αρχή. Ε, ε, επίσης ε, ανησυχώ για ορισμένες τροπολογίες και ορισμένες πτυχές της εκθέσεως του εισηγητή και γι' αυτό έχω υποβάλει τροπολογίες και το σύστημα αυτό δεν πρέπει να λειτουργεί μόνο σε λίγες χώρες και καλό θα ήταν να λάβουμε υπόψη μας ότι η οι νομικές διατάξεις για τα δικαστήρια διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Πρέπει να υπάρχει εφαρμογή και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καλή συνεργασία και γι' αυτό ε, συγχαίρω τον εισηγητή και τους ε, ε, συνεργάτες του. Ο κύριος Μέλο, για να ολοκληρώσει. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που παρενέβησαν στη συζήτηση αυτή και θα ήθελα για άλλη μια φορά να επαναλάβω τη θέλησή μου να φτάσουμε σε τροπολογίες συμβιβασμού και σε συμβιβασμούς γενικότερα κατά την μελλοντική ψηφοφορία. Νομίζω λοιπόν ότι η οδηγία αυτή έχει μεγάλη σημασία για την Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας και θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια έτσι ώστε να συμπεριλάβουμε τις τροπολογίες που δεν αλλοιώνουν το κανονιστικό και ρυθμιστικό πλαίσιο του κειμένου που θα ψηφιστεί στο σύνολό του. γιατί αυτό που έχει σημασία είναι να υπάρχει συνοχή, κανονιστική συνοχή. Νομίζω ότι έχουν συγκλίνει αρκετά οι θέσεις και αυτό αντικατοπτρίζεται και στις τροπολογίες όπου αναφερόμαστε στις ε, ανησυχίες και στα μελήματα των συναδέλφων Οπωσδήποτε η δικαιοσύνη είναι κάτι το υπερεθνικό και διακρατικό. Δεν ήθελα να επαναλάβω αυτά που είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα στην Ουάσιγκτον. Υπάρχουν πολλά στοιχεία σύγκλησης. Θα ήθελα να πω προς την κυρία Βέμπερ ότι όταν μιλάμε για αξι... αξιόπινες πράξεις έχει σημασία να γνωρίζουμε ποια είναι η εμβέλεια αυτών των αξιόπινων πράξεων. Είναι πτέσματα ή πλημελήματα. Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Στη χώρα μου δεν υπάρχει επαρκής ε, ορισμός των ε, πτεσμάτων, δηλαδή το, πνέσμα, το πτέσμα με συγχωρείτε, αλλιώς ορίζεται στην Πορτογαλία και αλλιώς στη Ρουμανία ή στη Γερμανία. Γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε να κάνουμε με ένα κείμενο το οποίο να μπορεί να μεταφερθεί στις 27 εσωτερικές ένομες τάξεις και υπό αυτή την οπτική γωνία θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την οδηγία. Δηλαδή να λάβουμε υπόψη την ε, ένομη τάξη των κρατών μελών. Ως προς τις προσφύγες θα πρέπει να δούμε πώς ορίζονται στο κράτος έκδοσης, στο κράτος συζήτησης και στο κράτος εκτέλεσης. Δηλαδή η δυνατότητα προσφυγής ορίζεται μόνο στο κράτος έκδοσης ή και στο κράτος συζήτησης, στο κράτος δηλαδή της ε, ακροαματικής διαδικασίας. Γιατί σε αυτή την περίπτωση τι θα ισχύσει και στο κράτος εφαρμογής, εκτέλεσης δηλαδή θα πρέπει να έχουμε ένα τυπικό ορθολογικό πλαίσιο, έτσι ώστε να μην ε, προβαίνουμε σε υπερβολικές τυποποιήσεις που οδηγούν στη μη εφαρμοσιμότητα της οδηγίας, γιατί τότε ε, αποσύρουμε την αποδοτικότητα μίας διάταξης. Και αυτό το βλέπουμε ιδιαίτερα στο νότο της Ευρώπης. Θα πρέπει να βρούμε μία εξισορροπημένη λύση ως προς τις ε, εγγύησεις των δικαιωμάτων, την εγγύηση των δικαιωμάτων των πολιτών. Να μιλάμε για δημόσιο συμφέρον και για, τα, για καταπολέμηση του εγκλήματος και ιδιαίτερα κατά πολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος που κατέχει δεσπόζουσα θέση πλέον. Γι' αυτό ακριβώς δεν θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα προσφυγής και στα δύο κράτη. Διαφορετικά εξουδετερώνουν την ιδέα. Θα πρέπει να υπάρχει αμοιβαία αναγνώριση. Αυτό το αναγνωρίσουμε και το κράτος ε, εκτέλεσης δεν θα πρέπει να τρέφει υποψίες ως προς το κράτος ε, συζήτησης. Έχει μεγάλη σημασία το δικαστήριο να αποφανθεί εκτιμώντας τα αποδεικτικά στοιχεία με βάση το νόμο και το δίκαιο έχουμε να κάνουμε με κράτη δικαίου. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Και γι' αυτό δεν θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα της διτής προσφυγής. Θα πρέπει να το διευκρινίσουμε. Ποιο δικαστήριο μπορεί να προσφύγει, το ένα και τα δύο ή πώς θα οριστεί. Εάν λοιπόν ένα φυσικό πρόσωπο πρέπει να μεταβεί από ένα ε, κράτος στο άλλο, θα πρέπει να είναι σίγουρο ότι δεν υπάρχει διαφορετική μεταχείριση. Οι σκέψεις σας είναι ίδιες με τις δικές μου. Αν θέλετε μπορούμε και να το συζητήσουμε και θα ήθελα να πω ότι έχει μεγάλη, έχουν μεγάλη σημασία οι τηλεφωνικές υποκλοπές και οι εγκρυπτό παρακολουθήσεις γενικότερα. Θα πρέπει να δούμε πώς ορίζεται το πλαίσιο από το κάθε κράτος μέλος. όλα αυτά θα πρέπει να τα έχουμε υπό απόλυτο έλεγχο. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και για τα όσα είπατε ως προς τη γενικότερη παρακολούθηση και τις υποκλοπές. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Επιτροπή και το Συμβούλιο για τις προσπάθειες που κατέβαλαν διότι αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε τι διαφορές υπάρχουν και μεταξύ ε, θεσμικών οργάνων. Γι' αυτό και προβάλλουμε τριμερή διάλογο για τέτοια θέματα ύψης της σημασίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Μέλλο. Ευχαριστώ και όλους τους συναδέρφους για τη συνεργασία. Ερχόμαστε στο τελευταίο σημείο της σημερινής μας ημερήσιας διάταξης που είναι το σημείο 7. Πρόκειται για τροποποίηση του κανονισμού περί καταλόγου τρίτων χωρών, υπήκο των οποίων υπόκειται στην υποχρέωση θεώρησης. Όπως θα θυμόσαστε ήδη στη συνεδρίαση της ΛΥΜΠΕ της 25ης Ιανουαρίου, στα πλαίσια της πρώτης ανταλλαγής απόψεων που είχαμε επί των τροπολογιών που είχαν καταθέσει οι ευρωβουλευτές του σχέδιου έκθεσης, ο εισηγητής, ο κύριος Ντίεθ Δεμέρα, ε, τέθηκαν ε, θέματα νομικά για το κατά πόσο υπάρχει αυτοματισμός εφόσον πρόκειται για επαναφορά της υποχρέωσης θεώρησης και είχαμε επίσης την τροπολογία 28 που έχουν υπογράψει διάφοροι ευρωβουλευτές και την τροπολογία 10 του εισηγητή. Ζητήσαμε λοιπόν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 Επειδή έχουμε λίγο χρόνο στη διάθεσή μας, θα είμαι σύντομος. Όπως είπατε και εσείς, πράγματι υπάρχουν δύο πτυχές στις ε, τροπολογίες 10 και 28 που εγείρουν νομικά ζητήματα. Και οι δύο τροπολογίες έχουν ως ε, στόχο να εισαγάγουν έναν πιο αποτελεσματικό μηχανισμό αμοιβαιότητα στις περιπτώσεις όπου τρίτη χώρα η οποία αναφέρεται στο παράρτημα 2 του κανονισμού 539 κάθετος 2001, μια χώρα δηλαδή ε, για την οποία δεν υπάρχει υποχρέωση θεώρησης, επιβάλλει υποχρέωση θεώρησης για υπηκόους κάποιας χώρας μέλους. Η νομική υπηρεσία όμως για να απαντήσει στο ερώτημά σας πρέπει να επενθυμίσει ότι ισχύει η αρχή της δοτής αρμοδιότητας και βάσει της αρχής αυτής τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν ελεύθερα να αποφασίζουν με ποιον ε, με ποιο τρόπο θα παίρνουν τις αποφάσεις τους, αλλά θα πρέπει να τηρήσουν τις διαδικασίες που προβλέπονται στη συνθήκη. Η υποχρέωση αυτή που απορρέει τόσο από το πνεύμα όσο και από τη διατύπωση και τη λογική των συνθήκων έχει επαναληφθεί ξανά και ξανά και από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σε μια σημαντική δικαστική απόφαση που ήταν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εναντίον Συμβουλίου που είχε να κάνει με τη λεγόμενη παράγωγη νομική βάση, ήταν μια περίπτωση για κύρωση κάποιων διατάξεων όσον αφορά την οδηγία για το άσυλο. Τότε λοιπόν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είπε ότι οι κανόνες που έχουν να κάνουν με τον τρόπο με τον οποίο τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα καταλήγουν σε απόφαση προβλέπονται από τις συνθήκες και συνεπώς δεν μπορούν τα κράτη-μέλη ή τα θεσμικά όργανα από μόνα τους να κάνουν ό,τι θέλουν. Η τροπολογία 10 αναφέρει μια διαδικασία για υιοθέτηση απόφυσης όσον αφορά την προσωρινή επαναφορά της υποχρέωσης θεώρησης για μια περίοδο 12 μηνών μέσω μιας κοινή νομοθετικής διαδικασίας. Η διαδικασία λήψης απόφασης δεν είναι το πρόβλημα. Όμως αυτό που είναι πρόβλημα είναι ότι η τροπολογία αυτή προβλέπει μια υποχρέωση για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για την υιοθέτηση μιας απόφασης όσον αφορά την επαναφορά υποχρέωσης θεώρησης. Υπενθυμίζουμε εδώ ότι το δικαίωμα της Επιτροπής για νομοθετική πρωτοβουλία είναι ένα πολύ βασικό στοιχείο στην διαθεσμική ισορροπία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι εκείνη η οποία προτείνει ποια στιγμή θα υποβάλει τέτοια νομοθετική πρόταση. Σύμφωνα λοιπόν με τις διατάξεις των συνθήκων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει περίπου αποκλειστικά το δικαίωμα της νομοθετικής πρωτοβουλίας. Συνεπώς, ε, βάζοντας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την υποχρέωση να υποβάλει νομοθετική πρόταση αυτόματα μετά από μια συγκεκριμένη κατάσταση, η τροπολογία 10 δεν σέβεται τα προνόμια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την νομοθετική πρωτοβουλία. Το δεύτερο ερώτημά σας τώρα έχει να κάνει κυρίως με την τροπολογία 28 και έχει να κάνει με ε, το κατά πόσο είναι σύμμορφη η πρόταση για τον μηχανισμό λήψης απόφασης. Ο μηχανισμός αυτός προβλέπει μία αυτόματη υιοθέτηση ε, πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκτός αν ρητά την έχουν απορρίψει το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Το πρόβλημα όμως με το κείμενο της τροπολογίας αυτής είναι ότι δεν αντιστοιχεί στην ισχύουσα διαδικασία βάσει του άρθρου 77 δύο των συνθήκων, δηλαδή την ε, κοινή νομοθετική διαδικασία, ούτε με καμιά άλλη προβλεπόμενη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Φαίνεται να προτείνει μια νέα διαδικασία, η οποία δεν προβλέπεται από τις συνθήκε. Σύμφωνα λοιπόν με την υπάρχουσα νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου μπορούμε να καταλήξουμε στο ότι εφόσον προσπαθεί να προβλέψει κάποιο είδους εναλλακτική διαδικασία, η τροπολογία 28 δεν, είναι, δεν συνάδει και δεν είναι σύμμορφη με τις ε, διατάξεις των συνθηκών. Όσον ε, αφορά λοιπόν τα προηγούμενα νομική υπηρεσία τονίζει ότι και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει αποφαθεί σχετικά με την παράγωγη ε, νομική βάση και άρα είμαστε μπροστά σε μια διαδικασία που δεν ε, είναι σύμμορφη με τις συνθήκες και άρα δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ε, ε, ισχύουσα. Και δεν μπορεί να είναι και δεσμευτική για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Συνεπώς, ε, κάποιο είδους αντιστραμμένος μηχανισμός ε, ψηφοφορίας που θα έχει σαν αποτέλεσμα να διαχωρίζει την ευθύνη για την πράξη από την εξουσία απόφασης για την πράξη, είναι κάτι που ε, μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν ε, συμμορφώνεται με τις συνθήκες. Είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρόεδρος, ο κύριος Διαθεμέρα, τώρα εισηγητής, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. θα κάνω ένα σχόλιο που έχει να κάνει με την γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας. Πέρα από την θέση μου, θέλω να σας προειδοποιήσω, να σας πω ότι η διάθεσή μου είναι επικοδομητική και συμφιλιωτική. Παρ' όλα αυτά, που θα ακούσετε σχετικά με την γνωμοδότηση τοπική υπηρεσία που λέει ότι η αναθεώρηση του κανονισμού 539 θα ενισχύσει την νομική ασφάλεια. Ωραία. Συμφωνώ ότι αυτό είναι ο στόχος της πρότασης. Σύμφωνα με τη συνθήκη και τον κώδικα για τις θεωρήσεις και του κανονισμού 810. Συνεπώς αυτό που θέλουμε είναι πράγματι να ε, διορθώσουμε την κατάσταση αυτή που επικρατεί όταν μια τρίτη χώρα αποφασίσει να επαναφέρει τις, ε, την υποχρέωση θεωρήσεων σε κάποια χώρα μέλος. Όμως έχουμε το θέμα της αμοιβαιότητας εδώ και η αμοιβαιότητα είναι το πιο σημαντικό στην πρόταση που μας απασχολεί σήμερα. Αυτό λοιπόν που θέλουμε είναι πιο αποτελεσματική αμοιβαιότητα. Και που να βασίζεται βέβαια στην αρχή της νομιμότητας. Η τροπολογία αριθμός 10, την οποία ε, αξιολογεί η Νομική Επιτροπή, λέει ότι μετά από διαβούλευση με το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος θα προτείνει την αμοιβαιότητα για 12 μήνες και βάση της κοινή νομοθετικής διαδικασία. Δεν θα σχολιάσω την τροπολογία αριθμός 28, γιατί αυτό είναι κάτι που μπορούν να κάνουν εκείνοι που την έχουν υποβάλει και την υποστηρίζουν. Πάντως εγώ δεν συμφωνώ με την τροπολογία 28. Και ανεξάρτητα με τον σεβασμό που έχω απέναντι σε όλους όσοι την συνυπογράφουν. Επανέρχομαι λοιπόν στην τροπολογία 10 και την γνωμοδότηση τη Νομική Επιτροπή. η νομική υπηρεσία μα παραδέχεται ότι πρόκειται για μια προσωρινή ρύθμιση. Κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι ένα πιο αποφασιστικό βήμα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα έστελνε ένα μήνυμα στην τρίτη χώρα η οποία μας επιβάλλει την υποχρέωση θεώρησης. Όσον αφορά τώρα τις γενικές παρατηρήσεις της νομικής υπηρεσίας, η τροπολογία μου 10 δεν ε, αντιβαίνει στο άρθρο 13, ούτε στο άρθρο 7 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γνώμη τους και γνώμη μου. Μέχρι τώρα η η γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας το μόνο που κάνει είναι ότι αναφέρει τα ήδη γνωστά έτσι όπως αναφέρονται στα δύο αυτά άρθρα, 13 και 7. Το σημείο 11 της έκθεσης λέει ότι το δικαστήριο είπε ξεκάθαρα ότι οι ρυθμίσεις που έχουν να κάνουν με τον τρόπο με τον οποίο τα θεσμικά όργανα λαμβάνουν τις αποφάσεις τους περιλαμβάνονται στις συνθήκες. και δεν μπορούν τα κράτη-μέλη ή τα θεσμικά όργανα να κάνουν από μόνο τους αυτό που θέλουμε. Είναι μια γενική παρατήρηση αυτή. Έπειτα το σημείο 12 για μένα είναι τόσο προφανές που δεν χρειάζεται κανένα σχόλιο. Το 13, 14 και 15 που έχουν να κάνουν με τις νομοθετικές ε, πράξεις το 288 και 289 που κάνουν διάκριση ανάμεσα στην ε, τακτική νομοθετική διαδικασία και τις έκτακτες Ούτε και αυτά τα σημεία χρειάζονται ιδιαίτερο σχόλιο. Μετά στην νομοδότηση μιλάει για τις κατεξουσιοδότηση πράξεις βάσει του άρθρου 209 της Συνθήκης Λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και το 291. Υπάρχει όμως και το σημείο 16, το οποίο λέει ρητά ότι για τις ε, καταξιδότηση ε, πράξεις και ιδίω για αυτές που το Συμβούλιο η συνθήκη λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν καθορίζει διαδικασίες, δεν καθορίζει διαδικαστικές διατάξεις. Έτσι λέει. Και συνεχίζω. Αναφέρει όμως ένα κανονισμό του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για να καθορίζονται οι γενικές αρχές που έχουν να κάνουν με τον έλεγχο που κάνουν τα κράτη-μέλη. Έλεγχο από τα κράτη-μέλη. Για θέματα... Για τι θέματα μιλάμε. Εδώ δεν είναι ένα θέμα το οποίο επιδέχεται ερμηνεία μιλάει για ελέγχους από τα κράτη-μέλη στις αρμοδιότητες της εκτελεστικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δηλαδή του Κοινοβουλίου, που έχει τη δυνατότητα ελέγχου και τα κράτη-μέλη. Αυτό λοιπόν που μας απασχολεί εδώ στην ουσία είναι το κατά πόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δηλαδή εγώ ο ηγητής σε σχέση με την τροπολογία 10, με τακτική νομοθετική διαδικασία μπορώ νόμιμα ή δεν μπορώ να υποβάλω την τροπολογία αυτή χωρίς να προσβάλλω το δικαίωμα νομοθετικής πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή είναι η ουσία του ζητήματος της τροπολογίας 10 και αυτό είναι ε, για το οποίο ζητήσαμε γνωμοδότηση από την νομική υπηρεσία μας. Όσον αφορά για το Β, η πρώτη ερώτηση απαντάει το, με το σημείο 18 που λέει ότι γιατί η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν μπορεί να υποβληθεί στην τακτική νομοθετική διαδικασία εφόσον η ίδια η πρόταση της Επιτροπής στο σημείο Γ λέει και διαβάζω ότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σε σχέση με την πρόταση αυτή θα αντιδράσουν με την τακτική νομοθετική διαδικασία. Έτσι λέει στο σημείο γάμα της πρότασής της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η διαδικασία λοιπόν για την υιοθέτηση μιας απόφασης επιβάλλει μια τροποποίηση των παραρτημάτων κανονισμός 539 που μιλάει για τις προσωρινές ρυθμίσεις και όλοι γνωρίζουμε και εσείς και εγώ ότι ο κανονισμός αυτός δεν είναι μόνιμος, έχει ήδη τροποποιηθεί 8-9 φορές. Είναι μικρής διάρκειας δηλαδή. Έπειτα, σημείο 20 της γνωμοδότησης, συμφωνώ. Σημεία 21, 22 και 23 δεν συμφωνώ κυρίως με το 24, όπου λέει το εξή λέει ότι για να υπάρξει απόλυτη υποχρέωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκειμένου να υποβάλει νομοθετική πρόταση ως ε, αυτόματη αντίδραση μετά από μια δεδομένη κατάσταση. Και λέει ότι η τροπολογία 10 δεν σέβεται το προνόμιο αυτό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εγώ δεν συμφωνώ. Και γιατί? Για τους εξής λόγους. Η πρόταση, δηλαδή η τροπολογία 10 του εισηγητή, μοιάζει πάρα πολύ με τη θέση της ίδιας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στις δύο περιπτώσεις η έκθεση αυτή μπορεί να συνοδεύεται από πρόταση, λέει η Επιτροπή. Θα προτείνει, λέει ο εισηγητής. Έπειτα και στις δύο περιπτώσεις μιλάμε για μια προσωρινή αποκατάσταση επαναφορά. Στο σημείο 19 της ε, γνωμοδότησης. Έπειτα η παράταση. Αναφέρεται η τροπολογία 10 και λέει ότι η παράταση αυτή εξαρτάται από το... Μάλλον δεν προκαταλαμβάνει το δικαίωμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προτείνει τροποποίηση του κανονισμού 539. Στη συνέχεια και στις δύο περιπτώσεις μιλάμε για αποφάσεις στις οποίες συμμετέχει και το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. 5. Στο δέλτα της τροπολογίας 10 λέει ότι η Επιτροπή εφόσον θεωρεί ότι πρέπει μπορεί χωρίς προηγούμενη έκθεση κλπ. κλπ. Εγώ καταλαβαίνω ότι με αυτό σέβομαι απόλυτα το δικαίωμα πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και η τροπολογία 10 λέει στο ε ότι δεν θα επηρεάσει το δικαίωμα της Επιτροπής να υποβάλει πρόταση τροποποίησης. Επαναλαμβάνω και πάλι ότι έτσι σέβομαι το δικαίωμα πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το δικαίωμα πρωτοβουλίας της Επιτροπής. Εβδόμο, τροπολογία 10 και η θέση της Κομισιόν μιλάνε για την κοινή νομοθετική διαδικασία. Άρα και εγώ το κάνω. Και δύο μιλάμε για την τακτική νομοθετική διαδικασία. Κατά τα άλλα, η πλειοψηφική θέση του Συμβουλίου λέει στο γάμα ότι 90 μέρες μετά ε, την λήψη και κατά τη διάρκεια έξι μηνών μετά από την ημερομηνία δημοσίευσης, δηλαδή η ανακοίνωση έχει δύο δυνατότητες. Η μία είναι ότι το Συμβούλιο λέει στην Επιτροπή, εσείς έχετε δύο εναλλακτικέ. Αυτό λέει το Συμβούλιο στην Επιτροπή. Τη λέει τι πρέπει να κάνει, τη δείχνει το δρόμο. Τη λέει ένα από τα δύο πράγματα θα κάνει. Ή που θα δεχτεί απόφαση εφαρμογής της άρσης ή που θα υποβάλεις έκθεση αξιολόγησης. Και στις δύο περιπτώσεις, δηλαδή, το Συμβούλιο δεν αφήνει την Επιτροπή να κάνει ό,τι θέλει. Της λέει, έχεις αυτές τις δύο επιλογές. Δύο, όχι παραπάνω. Πού είναι εδώ λοιπόν το δικαίωμα πρωτοβουλίας που θέλουμε να προστατεύσουμε της Επιτροπής. Ενώ πρόκειται για υποχρέωση βλέπετε. Το Συμβούλιο εδώ υποχρεώνει την Επιτροπή της, εκφράζει την απόλυτη υποχρέωση που έχει για νομοθετική πρόταση. Ενώ η δικιά μου η τροπολογία 10 δεν επιβάλλει τέτοια πράγματα. Συνεπώς, δεν λέω ότι έχω καταλήξει, παραμένω ανοιχτός στις διαπραγματεύσεις, να συζητήσουμε όλες τις νομικές και μη νομικές λεπτομέρειες. Θέλω να συζητήσω με τους συναδέρφους αλλά και με την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Και ευχαριστώ πολύ την νομική υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την δουλειά της που είναι πάντα αναγκαία προκειμένου να μας βοηθήσει στο νομοθετικό μας έργο. Και προτείνω να καταλήξουμε σε μια συμφωνία με τους σκιώδεις εισηγητές και όσους υπέβαλαν τροπολογίες για να βρούμε μια λύση στο μοναδικό θέμα που μένει να λύσουμε σε αυτή την υπόθεση, που είναι το θέμα της αμοιβαιότητας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Δίας Δεμέρα. Έχω τρεις ομιλητές, τρεις συναδέλφους που θέλουν να επέμβουν, τέσσερις. Θέλω όμως να σας πω ότι έχουμε έξι λεπτά ακόμη και ξέρω ότι θα πρέπει να είστε σύντομοι διότι ε, επειδή το προηγούμενο θέμα ε, μακρηγόρησε περισσότερο πρέπει να σας παρακαλέσω να είστε πάρα πολύ σύντομοι. Η κυρία Φαγιών. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη γιατί έχουμε συνέχεια και μια συνεδρίαση. Θέλω να ευχαριστήσω τους εισηγητές, διότι αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε εδώ είναι να βελτιώσουμε τον ισχύοντα μηχανισμό αμοιβαιότητος για να μπορέσει να είναι και λειτουργικός και νόμιμος και χωρίς να αποκλίνουμε από τη συμφωνία, γι' αυτό και ευχαρίστω θα συζητήσω για το πώς μπορούμε να δώσουμε δυνατότητα σε όλα τα κράτη-μέλη να ε, αντιδράσουν διότι ο μηχανισμός αυτός δεν είναι ικανοποιητικό και στον Καναδά παραδείγματο χάρη τα κράτη-μέλη δεν έδειξαν ε, την, ε, ε, την αλληλεγγύη που έπρεπε. Πρέπει λοιπόν να καταρτήσουμε ένα μηχανισμό ο οποίος θα προστατεύσει όλες τις χώρες και όλους τους πολίτες. Αντιλαμβάνομαι ότι τα περισσότερα κράτη-μέλη είναι ενάντια στην λύση ε, του να παρουσιάζει αυτομάτως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μία αίτηση θεωρήσεως για την είσοδο από τρίτη χώρα. Αυτό σύμφωνα με την ε, νομική γνωμοδότηση που ακούσαμε σήμερα και θα πρέπει να βρούμε τη σωστή διατύπωση, να προσαρμόσουμε και το δικό μας κείμενο και ίσως θα πρέπει να βρούμε κάποια λύση με την οποία θα μπορέσουμε να πιέσουμε περισσότερο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταρχήν να κάνει ό,τι μπορεί για να άρει τις υποχρεώσεις ε, θεωρήσεως και ε, να προτείνει τις προϋποθέσεις ε, θεωρήσεως στα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αιτιολογήσει ε, εάν δεν αποφασίσει να προχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Και είπατε ότι στην όλη αυτή τη διαδικασία το Κοινοβούλιο θα πρέπει να ενημερώνεται επί των αναγκαίων μέτρων. Πρέπει να πω ότι ο μηχανισμός αμοιβαιότητος δεν εμποδίζει να εφαρμοστούν και άλλα μέτρα για να υπάρχει ε, διακίνηση χωρίς θεωρήσεις, ε, χωρίς θεωρήσεις σύμφωνα με τις ε, διατάξεις των συνθήκων. Οπότε εγώ θα ήθελα να ξέρω ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο να βελτιώσουμε τη διατύπωσή μας και να έχουμε ικανοποιητικές λύσεις για όλους τους συναδέλφους. Ο κύριος Σαλβάρο. Ευχαριστώ κύριε ε, Πρόεδρε, ε, θα μπορούσαμε ίσως και να ψηφίσουμε ε, και να έχουμε ίσως και μία πλειοψηφία. Θέλω να ευχαριστήσω όμως και την Νομική Επιτροπή, γιατί δεν είναι τόσο εύκολο να γνωμοδοτήσεις το θέμα αυτό το οποίο πέραν νομικού είναι και πάρα πολύ πολιτικό θέμα. Είναι όμως θέματα τα οποία πρέπει να αξιολογήσουμε και να δούμε πώς θα προχωρήσουμε διότι διαμέσου των ετών έχω δει καλές τροπολογίες, κακές τροπολογίες και ανόητες τροπολογίες. Πιστεύω λοιπόν ότι στο σημείο αυτή, αυτή δεν είναι και πολύ πολιτικοποιημένη αλλά και σημαντική τροπολογία για να κατανοήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη που ε, ρωτούν είμαστε ισότιμοι. Όταν μιλάμε για τρίτες χώρες, ε, έχω κάνει και εγώ μία ε, μια τροπολογία, την τροπολογία 30, 29, ε, όπου λέγω ότι δεν υπάρχει προηγνούμενο από το γεγονός ότι δεν υπάρχει μια τροποποίηση η οποία να έχει υιοθετηθεί προηγουμένως, αλλά η τροπολογία 28 εισάγει έναν μηχανισμό αυτοματισμού που ε, ε, προέρχεται και απορρέει κατευθείαν από το six pack, από το σύνολο των έξι ε, οδηγιών το 1173, 75 και 76 ε, και υιοθετήθηκαν και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από την Επιτροπή και από το Συμβούλιο προ λίγων μηνών και ε, τα τρία λοιπόν θεσμικά όργανα συνένεσαν και τελικώς είπαμε ότι ο αυτοματισμός της αντιστρόφου πλειοψηφίας δεν είναι δεδομένο και χρειάζεται γνωμοδότηση της ε, νομικής ε, επιτροπής. Παρ' όλα αυτά υπερψηφίστηκε ε, και ο αυτοματισμός και αυτό τώρα προτείνει η διακομματική μας τροπολογία. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω ποια είναι η αντίδραση στο σημείο αυτό, διότι στο παρελθόν ο κύριος Μπαρόζο είχε πει ότι είναι ένα ποιοτικό βήμα προς τα εμπρός και ο κύριος Βούζεκ είχε μιλήσει ε, για ένα ισχυρό όπλο και οι, ε, οι κυρώσεις από τα κράτη-μέλη πρέπει να είναι ε, πιο αυτόματες. Ο κύριος Βαν είπε ότι είναι ευτυχής με τα επιτέχματα αυτά και πολλοί άλλοι είχαν ακολουθήσει ακριβώς το σημείο αυτό το οποίο αμφισβητούμε τώρα. Μπορώ να δεχθώ λοιπόν κριτικές σε πολιτικό επίπεδο, αλλά για ένα θέμα το οποίο έχει ε, ε, υπερψηφιστεί ε, και ένα μηχανισμό ο οποίος υπερψηφίστηκε εδώ και μήνες δεν κατανοώ την κατάσταση. Λοιπόν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να στηρίξει τους συναδέλφους στα άλλα κράτη-μέρη εφόσον το Συμβούλιο δεν ενδιαφέρεται να λύσει το πρόβλημα. Η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Πολωνία, η Τσεχία και πολλές άλλες χώρες έχουν πιέσει πολλές φορές για αμοιβαιότητα. Τα άλλα κράτη όμως τις αγνόησαν και πιστεύω ότι όπως και το σύνολο των έξι οδηγιών θα πρέπει και τώρα να εξασφαλίσουμε έναν μυθό μηχανισμό αμοιβαιότητος που να βαφίζεται στην αλληλεγγύη ακόμη και αν δεν είναι απόλυτα σωστό θα ήθελα να μας προσάγει στο δικαστήριο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφόσον θα το έχουμε αποφασίσει και ας έρθουν να μας πούν ότι δεν χρειάζεται αυτός ο αυτοματισμός και ότι δεν ενεργήσαμε σωστά. Εάν λοιπόν η Επιτροπή θέλει να μας ε, αφισβητήσει ευχαρίστως να φτάσουμε στα άκρα. Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπε ο κύριος ε, Άλβαρο και εγώ έχω συγκεκριμένες θέσεις ως προς τις τροπολογίες. Νομίζω ότι μπορούμε να βελτιώσουμε αυτή την επίμαχη τροπολογία όπως είπε και ο συνάδελφος ε, Άλβαρο, άλλοι θα αρνηθούν αυτή τη, τη σημασία αυτού του θέματος. Εδώ και τρία χρόνια που βρίσκομαι σε αυτή την Επιτροπή, ακούω διάφορες επικρίσεις για υποχρεώσεις, αμοιβέ υποχρεώσεις, καθήκοντα και δικαιώματα. Υπάρχουν όμως πολίτες πρώτης και δεύτερης κατηγορίες σε σχέση με τρίτες χώρες. Ποια είναι η κανονικότητα, ποιος είναι ο δρόμος για να τα καταφέρουμε έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να αρχίσει να διαπραγματεύεται αυτό το πλαίσιο. Γιατί μερικοί είναι πιο Ευρωπαίοι από τους άλλους. Η κυρία Τανόκα. Και εγώ θα ήθελα να πω λίγα ε, λόγια για την τροπολογία αυτή την 28. Νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε μια νέα διατύπωση η οποία να προσδώσει έναν αυτοματισμό για όλα τα κράτη-μέλη. Ο Αλεξάνδερ θέλει να κρατήσει την ίδια διατύπωση. Θα το συζητήσουμε, αλλά υποστηρίζουμε την ιδέα αυτή. Δηλαδή να έχουμε μία συνεπή θέση σε σχέση με αυτόν τον αυτοματισμό. Η νομική υπηρεσία έχει κάτι να προσθέσει. Πολύ σύντομα. Δύο σχόλια θα ήθελα να υποβάλω. Καταλαβαίνουμε ότι ο στόχος είναι να φτάσουμε σε έναν πιο αποδοτικό μηχανισμό αμοιβαιότητας για να απαντήσω στον εισηγητή. Γιατί αυτό προσπαθούμε να εκφράσουμε είναι το εξής. Αυτή η υποχρέωση στο C της τροπολογίας σας 5 δεν φαίνεται κατά τη δική μας άποψη συνεπής με το γράμμα των συνθήκων. Αναγνωρίζουμε όμως ότι η διατύπωση της παραγράφου Δέλτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο δηλαδή να χρησιμοποιηθεί και για την παράγραφο C, για το μικρό γάμα, για να επιληθεί το ζήτημα. Και κάτι άλλο. Γνωρίζω ότι ενδεχομένως έχει επέλθει συμφωνία μεταξύ κρατών μελών στο Συμβούλιο. Εμείς λάβαμε υπόψη τη νομική πλευρά δεν ξέρω κατά πόσο το Συμβούλιο θα συμβαδίσει. Ε, δηλαδή, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η νομική ακαιρεότητα του εγχείρηματος. Και ακόμα και αν είχαμε ορισμένα προηγούμενα, θα πρέπει να επισύρουμε την προσοχή και ως προς τα μέτρα εκτέλεσης δυνάμει του 291 στον κανονισμό του Συμβουλίου προσπαθούμε να σας δώσουμε άλλες πληροφορίες ως εναλλακτικές και γι' αυτό προχωρήσαμε λίγο παραπέρα. Αλλά το θέμα είναι δικό σας. Ο κύριος Δίας Δεμέρα θέλει κάτι να προσθέσει. Θέλετε να προσθέσετε κάτι, όχι. Ε, έχω καταγράψει τα όσα είπαν οι συνάδελφοι και η νομική υπηρεσία και μαζί με τους σκιώδεις θα δούμε τι δρόμο θα ακολουθήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ για σήμερα το απόγευμα, για τη συνεργασία σας. Θα συνεχίσουμε αύριο το πρωί στις 9 η ώρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα.